Παρακαλώ, αν θέλετε καθίστε. Συνεχίζουμε την σύνοδό μας. Σημείο 10 της ημερησίας διάταξης. Σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά. Τη 9 του μηνό ε, ανατέθηκε η, αυτή, η έκθεση αυτή στην κυρία Ντότζ. Σήμερα θα ακούσουμε την παρουσίαση από πλευρά τη Κομισιόν και μετά βέβαια θα συζητήσουμε το θέμα. Εκ μέρους της Κομισιόν, ποιος είναι εδώ? Many thanks, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν σας ε, παρουσιάσω την πρόταση για τη δεύτερη τροποποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου στο Κάτεγατ, ε, τη Βόρεια Θάλασσα και τον Ατλαντικό, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το ιστορικό. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης ισχύει από το 2008. Η απόδοση των μέτρων διαχείρισης του σχεδίου αξιολογήθηκε το 2011 από, τις, από την ε, ISIS και την ε, ε, Επιστημονική Επιτροπή Αλίας. Αυτή η αξιολόγηση εντόπισε συγκεκριμένες αδυναμίες ε, μεταξύ αυτών στο σχεδιασμό του κανονισμού και στην εφαρμογή του. Η διαδικασία αξιολόγησης ήταν δημόσια και συμμετείχαν τα περιφερειακά συμβούλια, οι ενδιαφερόμενοι και εκπρόσωποι των κρατών μελών. Επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης η Κομισιόν συζήτησε με τους εμπλεκομένους ε, τη δυνατότητα τροποποίησης της διαχείρισης των μέλων. Συμφωνήθηκε το σχέδιο που ισχύει να αντικατασταθεί από ένα μεικτό σχέδιο διαχείρισης σύμφωνα με την πολιτική αναδιάρθρωση της αλληλευτικής πολιτικής της Κομισιόν. Η... Τα μεικτά συστήματα είναι καινούρια προσέγγιση το επιστημονικό εργαλείο, τα επιστημονικά εργαλεία γι' αυτό, το λόγο, τα επιστημονικά εργαλεία που τα υποστηρίζουν δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Γι' αυτό το λόγο, πριν το 2014 δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτά τα μεικτά σχέδια να αρχίσουν να υιοθετούνται από την Κομισιόν. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν στο ισχύον ε, σχέδιο. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν προτείνει ένα, μια τροποποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες που ακούστηκαν από τα ΡΑΚ, από τα κράτη-μέλη και από την ε, επιστημονική αξιολόγηση που έγινε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εξ αρχής ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πλήρης αναθεώρηση του σχεδίου. Δεν πρόκειται να επιλύσει όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα χρειάζονται με καλύτερη αξιολόγηση αντικτύπου, και κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό στο χρόνο που μας είχε διατεθεί προκειμένου να επιλύσουμε τα βασικά ε, προβλήματα. Να σας δώσω μερικές λεπτομέρειες, αλλά πιο πριν θα σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν θα πρέπει να, ε, ε να, ε, ε, είναι, να θεωρηθεί ότι είναι ίδια με την πρόταση ευθυγράμμισης που υποβλήθηκε στην αρχή του χρόνου προκειμένου να τροποποιηθεί το ισχύον σχέδιο, προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι απαραίτητες τροπολογίες, ε, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία, η ισχύουσα νομοθεσία με την συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή τη στιγμή και στο στο συμβούλιο, συγγνώμη, στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο έχουμε δύο προτάσεις τροποποίησης του ε, σχεδίου για τον ε, ε, μία είναι η πρόταση για την ευθυγράμμιση και μία είναι αυτή που συζητούμε σήμερα. Περνάμε στην ουσία της πρότασης που σας, προτείνουμε, που σας ε, παρουσιάζουμε σήμερα. Η... Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στην, τροπολο... στην τροποποίηση του άρθρου 4 του ισχύοντος κανονισμού. Αυτή η τροπολογία εισάγει την ε, απέτηση χρήσης της ίδιας μεθόδου υπολογισμού της ε, αλλιευτικής προσπάθειας ε, με τη μέθοδο που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη για, για τον υπολογισμό των baselines για την αλλιευτική προσπάθεια. Δεν αλλάζουμε την ίδια τη μέθοδο, απλά διευκρινίζουμε ποια μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται. Μια άλλη σημαντική τροποποίηση αφορά το άρθρο 9 του ισχύοντος κανονισμού. Η τροπολογία προτείνει μια διαδικασία για τον καθορισμό των ΤΑΚ απουσία των πληροφοριών που χρειάζονται για να εφαρμόσουμε τους συνήθεις κανόνες. Ε, σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε ανεπαρκή πληροφορίες, πληροφόρηση. το σχέδιο προτείνει αυτόματη μείωση 25% στο στατά και στην αλληλευτική προσπάθεια. Ε, αυτό ήταν ένα κανό ο οποίο είχε σκοπό να εφαρμοστεί μόνο, σε κατεξε... Πλην όμω στο Κάτεγα, στην Ιρλανδική θάλασσα και στην Δυτική Σκοτία, αυτή η κατεξέλιξη εφαρμογή έγινε τελικά συνήθι ο ισχύον κανόνας αν δεν τροποποιηθεί θα οδηγήσει μέσα σε μερικά χρόνια στην, στο κλείσιμο πρακτικά όχι μόνο της αλίας του γάτου αλλά και άλλων αλλιευμάτων που χρησιμοποιούν ε, τους τα ίδια λευτικά εργαλεία. Αυτό ενδεχομένως δεν είναι επιθυμητό σε όλες τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ο γάτος αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα των μεικτών αλλευμάτων. Σημαντικό λοιπόν είναι να τροποποιήσουμε τον κανόνα αυτό έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες ε, που αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ε, να επιτρέψουμε δηλαδή μεγαλύτερη ευελιξία. Η τροπολογία είναι, φαίνεται ίσως λίγο περίπλοκη, αλλά έχει ως στόχο να υιοθετήσουμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα μιας κατά περίπτωση αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα. Με αυτή την τροπολογία αποφεύγουμε αυτή την αυτόματη μείωση του 25% στα ΤΑΚ ή στην αλλιευτική προσπάθεια. Μια άλλη τροπολογία αφορά το άρθρο 11 της ισχύουσας νομοθεσίας. αποκλεισμό δηλαδή ε, σκαφών. Ε, κατόπιν αιτήματος της, ε, του τομέα, του κλάδου, η, ο αποκλεισμό ε, των ε, σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 11 αποδεχθήκαμε ότι είναι πολύ περίπλοκος. Η πρότασή μας απλοποιεί αυτή την, αυτό τον αποκλεισμό. Οπότε θεωρούμε ότι η τροπολογία προτείνουμε θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου περισσότερα σκάφη θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτό αυτή την εξαίρεση ε, και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και θα αυξηθεί η χρήση πιο επιλεκτικών εργαλείων. Θα ε, προωθήσουμε λοιπόν περισσότερα επιλεκτικά, εργαλεία, περισσότερα επιλεκτικά εργαλεία και θα αποφύγουμε επίσης να αλλιεύουμε εκεί που υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις γάδων. Ε, σε αυτή την τροπολογία επίσης προβλέπουμε ε, τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν ε, σε αλίευση για τα οποία έχουμε πλήρη περιπληροφόρηση μπορούν να αποκλείονται υπό την προϋπόθεση ότι ε, βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του τάκτους. Η παρούσα αυτή η τροποποίηση του άρθρου 11 ε, ε, όπως και η τροποποίηση του άρθρου 9 δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισμό των αιτήσεων, ε, της αιτήσεως αλευτικής προσπάθειας. Η Κομισιόν ε, ρώτησε, έχει ζητήσει την Επιστημονική Επιτροπή Αλίας να μας ε, πει αν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες καθορισμού των τάκετ της αλληλευτικής προσπάθειας σε τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή όταν δεν έχουμε αρκετά επιστημονικά δεδομένα. Επιπλέον, σε αυτή την τροπολογία δυνα... Ε, το Συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει κάθε χρόνο αν θα εφαρμόζει περαιτέρω μειώσεις της ε, αλληλευτικής προσπάθεια. Το 2013 σας πω ότι θα γίνει η πεντηκοστή προσπάθεια τη αλληλευτικής προσπάθεια σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης στις τρεις από τις τέσσερις περιοχές που καλύπτονται από το σχέδιο η μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας για τα βασικά εργαλεία αλληλεύσης ε, του γάδου ε, είναι 25% κάθε χρόνο από την υιοθέτηση του σχεδίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις ε, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στους εμπλεκομένους. Ανοίγουμε λοιπόν τη δυνατότητα το Συμβούλιο να αποφασίζει ετησίως αν θα εφαρμόσει περαιτέρω μειώσεις ε, στην αλευτική προσπάθεια κάθε φορά. Στην τροποποίηση του άρθρου 14 τώρα. Υπογραμμίζουμε την ε, υποχρέωση ο πλευράς των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν το θέμα ε, των απορρίψεων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υψηλού επίπεδου απορρίψεων. Υπάρχουν μερικές περιοχές όπου ε, έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα απορρίψεων γάδου. Συνεπώς τα κρατη μελη είναι σημαντικό να συνεχίσουν να παίρνουν τα μέτρα που θα βοηθήσουν να αποφύγουμε τέτοιου είδου ε, επίπεδα απορρίψεων. Η πρόταση επίσης αναφέρει τα επίπεδα ελέγχου ε, για τα σκάφη με βάση την ε, στρατηγική αξιολόγηση κινδύνου. Πρέπει δηλαδή να έχουμε ε, μια στρατηγική αξιολόγηση κινδύνου και με βάση αυτή να κάνουμε τους ελέγχους. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις κομισιών, σύμφωνα με την νομοθετική δομή της Συνθήκης Αβώνας, η πρόταση δίνει την αρμοδιότητα στην Κομισιόν να ε, υιοθετεί εφαρμοστικές πράξεις για τη διαδικασία ενημέρωσης ε, και μετάδοση πληροφοριών στην Κομισιόν δεν έχουμε προβλέψει για να αποφύγουμε μπλοκάσμα ε, ε, μεταξύ των οργάνων δεν έχουμε προβλέψει κατεξιοδότηση πράξης. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να υιοθετήσουμε κάποιες εξειδόξη τη πράξη για να απλοποιηθεί η διαδικασία, υπό την προπόθεση βέβαια ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν. Τέλος να πω ότι η υιοθέτηση αυτής της πρότασης είναι ιδιαίτερα πήγουσα. τουλάχιστον αυτό λένε τα κράτη-μέλη και οι εμπλεκόμενοι φορείς του κλάδου. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι η πρότασή μας έχει υποστηριχθεί εν γέννη και από τα κράτη-μέλη και από τον κλάδο. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την κυρία Ντότς που, ε, έχει, που κάλεσε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής του 8 Οκτωβρίου τους αντιπροσώπους των ΡΑΚΣ. Και τα δύο ΡΑΚΣ που προσκλήθηκαν ε, υποστήριξαν ε, την πρότασή μας και είναι προφανές ότι είναι πήγον να υιοθετηθεί σύντομα. Ο φάκελο αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει, επίση προχωράει γρήγορα στο Συμβούλιο. Έχει ήδη συζητηθεί δύο φορέ και, έχει προβλεφθεί άλλη μια συζήτησή του αυτή τη βδομάδα. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε την πρότασή μα, την παρουσίασή μου και αναμένω μια επικοδομητική συνεργασία με εσά. Άμα θέλετε μπορώ να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή που με όρισε ως εισηγήτρια για την ε, αναθεώρηση ε, της σύστασης μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα θέματα γάδου γιατί σε ό,τι αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιρλανδία και τι Καναδικές χώρε γιατί είναι κάθε μελιώδες. Πρέπει βέβαια να έχουμε αυτή την ε, έκθεση ευθυγράμμιση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, αλλά δεν πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να γίνεται σύγχυση στην Επιτροπή ανάμεσα στα δύο. Μπορούμε να έχουμε την έκθεση ευθυγράμμιση και εκ αυτή την ιδιαίτερη έκθεση που ουσιαστικά τροποποιεί το σχέδιο. Δυστυχώς ε, η έκθεση ευθυγράμμισης θα αποτελέσει αντικείμενο διαθεσμικής συζήτησης και μπλοκαρίσματος, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ελπίζω ότι με ούριο άνεμο και με συνεργασία Συμβουλίου και Επιτροπής θα μπορέσουμε στην Επιτροπή αυτή να προχωρήσουμε την έκθεση αυτή σχετικά γρήγορα. Θα ήθελα να πω αυτή εξ αρχής ότι μία από τις ε, πτυχές ε, της ε, έκθεση αυτή που προέκυψε πολύ έντονα αποτελεί ένα μάθημα για όλους μας σε σχέση με τις ε, εργασίες μας. Όπως ε, είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αυτή η έκθεση είναι μετά από μια αξιολόγηση που έγινε το 2011 που εντόπισε συγκεκριμένες σημαντικές αδυναμίες και στον κανονισμό και στη σύνταξη του κανονισμού και στην εφαρμογή του. Υποθέτω ότι κάτι που για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας έχει προκύψει με πολύ μεγάλη συνεργασία από τους εμπλεκόμενους φορείς και από τα περιφερειακά συμβούλια και αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά επίγοντα και κέρια στον τομέα, θα πρέπει πάντα να συνεργαζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ακριβώς όπως είπα και προσώπων ε, του τομέα αυτού από τις κατατόπου χώρες. Δεν αποτελεί μια αντικατάσταση του σχεδίου, αλλά μια, ένα καλύτερο φινίρισμά του, όπως θα έλεγα, προτού το υιοθετήσουμε, προτού υιοθετήσουμε που θα θέλαμε να δούμε νομίζω όλοι εμείς ένα μεικτό σχέδιο, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Την περασμένη εβδομάδα μια ε, επιτροπή ε, αλλιέων από τη Βόρεια Ιρλανδία ταξίδεψαν στην Νορβηγία. Μίλησα μαζί του Σαββατοκύριακο και μπορούσαμε να τα πολύ ευχάριστα νέα και πρέπει να τα γνωρίζουμε τα καλά νέα, γιατί ορισμένε φορέ είναι δύσκολο να βρούμε και καλά νέα. Το σημαντικό ήταν η ανάπτυξη των αποθεμάτων γάδου στην Βερίγκια θάλασσα όπου ενδεχομένω του χρόνου περιμένουν πάνω από ένα εκατομμύριο τόνων, τόνων, που είναι πολύ σημαντική αύξηση. Πράγμα το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και δεν θα πρέπει να το ελαχιστοποιούμε. Δεν πρόκειται να εξετάσω μία προς μία τις ε, τροπολογίες. Θα ήθελα όμως να εκφράσω κάποιες σκέψεις για το θέμα. Όπως είπα, αισθάνομαι ότι είναι πραγματικά ένας ε, σημαντικός, ένας ακρογωνιαίος λίθος. Είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιου είδους ε, σημαντικούς, ε, σημαντικούς σταθμούς προχωρώντας στην αναθεώρηση αυτού του μακροπρόθεσμου σχεδίου. Έχουμε ήδη το άρθρο 4 που αφορά στην διαχείριση των προσπαθειών. Ξέρουμε ότι πολύ σημαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί από το 2009 αλλά που όμως δεν υπήρξαν αποτελεσματικές. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν λογικό να αποσαφηνίσουμε τους κανόνες σε σχέση με τα κράτη-μέλη, τις ε, ε γραμμές ε, ε, προσπαθειών. Το άρθρο 9 νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί και έχει προκαλέσει πολλές ερωτήσεις. Το 2008 ένα από τα σημαντικά ε, σχέδια τα οποία υπήρχαν, οι διαφορές, είναι να αλλάξει τα θέματα αποτελεσματικότητας στην αλίευση ε, γάδου και βακαλάου. Η άμεση υποκατάσταση κατά 25 των υπάρχει στο άρθρο 9 και ε, εξετάζει την κατάσταση των ΤΑΚ αναπερίπτωση. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό και εισάγει μια ευελιξία που όλοι ε, τις οποίες όλοι υπεραμεινόμεθα σε αυτή την Επιτροπή και το ζητάει και ο τομέας της Αλίας. Το άρθρο 11 εξετάζει τις εξαιρέσεις για τα σκάφη εκείνα που αλλιεύουν αμελητές ποσότητες ε, βακαλάου και είναι στον απόϊχο λογικών ε, διαφορών και έχει τρόπο ακριβώς και ευθυγραμμίζεται στο να επιλέγουν τα σκάφη αντίστοιχο εξοπλισμό. Άρα και πάλι είναι σωστό αυτό γιατί εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία στο σχέδιο αυτό. Είναι καλό και ακριβώς ε, μας βοηθά να μην πηγαίνουμε κάθε φορά να ανακαλύπτουμε τον τροχό, πάνω να σωστά πράγματα. Οι ε, εξαιρεσει για πλήρως πιστοποιημένες αλλιεύματα ξέρουμε ότι όλα τα αλλιεύματα συνοδεύονται με κάποιε συγκεκριμένε ε, ποσοστώσει. Υπάρχουν λοιπόν για κάθε τύπου σκάφου. Όμως, δεν θα ήθελα να, βλέπ, να δω μια διαχείριση των ποστόσεων εκτός αυτής που προβλέπεται ένα κράτος μέλος. Πρέπει να το δούμε, νομίζω, πιο λεπτομερώς, γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ε, απόπειρες ε, να υπονομευθεί αυτή η συγκεκριμένη αρχή. Η πρόταση για το άρθρο 13 που ε, εισάγει τις απαιτήσεις του 10% ποσόστος αλλιευμάτων είναι ένα προσδεκτό βήμα που θα μειώσει και τις απορρίψεις βακαλάου. Το άρθρο 14 ενισχύει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να μειώσουν τις απορρέψεις. Και όπως το είδαμε και στην ε, ε, ανάπτυξη εξαιρετικά εξειδικευμένου εξοπλισμού, ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει μια επικάλυψη μεταξύ αυτών των δύο μηχανισμών πρέπει να εισάγουμε, να ενθαρρύνουμε την επίτευξη των στόχων αυτών και ούτε η Κομισιόν, ούτε και τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν ε, λεπτομερείς οδηγίες σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς που θα πρέπει να ε, υπάρχουν πάνω στα σκάφη, αρκεί να μπορούν να καλύψουν ε, και να τεκμηριώνουν την μείωση των απορρίψεων. Θα συναντηθώ με την με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής και με κάποιους άλλους εκπροσώπους που μου ζήτησαν να με συναντήσουν. Εάν υπάρχουν και μέλη της Επιτροπής αυτής που έχουν ισχυρέ απόψεις πάνω στο θέμα και που θα ήθελαν να το συζητήσουν, να συζητήσουν συγκεκριμένη αυτή η έκθεση λεπτομερώς, είμαι στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και πραγματικά είναι ευπρόσδεκτη η συμβολή σας. Θα είναι πολύτιμη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά ε, τον, τους, ε, τους φιλοξενούμενους μας ε, Τώρα θα δώσω το λόγο στους, στους, στα μέλη μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω το Ευρωπαϊκό Κονσόρτιο για την Ανατολική Σκοτία. Ιδιαίτερα, ενώ, ιδιαίτερα καθώς συζητάμε ένα σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τα αποθέματα γάδου στην Δυτική Σκοτία και να ευχαριστήσω και την Diane Dodge για την παρουσίασή της. Έχω κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως η συγγήτρια θα μπορούσε να με βοηθήσει στην αποσαφήνισή τους. Φυσικά με χαρά άκουσα για την έλλειψη ελαστικότητας στις περικοπές 25% και ότι αυτό θα αλλάξει σύμφωνα με το άρθρο 9, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις μία-μία. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Θα καθυστερήσει την όλη διαδικασία, διότι χρειάζεστε επιστημονική συμβουλή, χρειάζεστε διαπραγματεύσεις στην εκάστοτε περίπτωση για το πώς θα προσεγγίσουμε αυτήν την νέα ελαστικότερη προσέγγιση για την ανάκαμψη του γάδου. Μετά θα απαιτήσει διαδικασία συναπόφασης. Το Κοινοβούλιο θα έχει κάποιο ρόλο. Θα συμμετέχει, διότι η διαδικασία είναι πολύ αργή. Επίσης, έχουμε δει πολιετή σχέδια τα οποία το Συμβούλιο τα δυσχεραίνει όλο ένα και περισσότερο. Το σχέδιο του κυρίου Γκάλαχερ για το Σαφρίδι ήταν ένα από αυτά. Εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο από την πρώτη ανάγνωση, αλλά τώρα έχει φτάσει σε αδιέξοδο και αυτό από το Συμβούλιο. Και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μας λέει ότι χαίρονται πάρα πολύ για αυτό το σχέδιο ανάκαμψης του γάδου. Αυτό είναι καλό. Αλλά θα μπορούσατε, Επιτροπή, να μας πείτε τι άλλαξε στη στάση αυτή και για την εφαρμογή του των πολιετών σχεδίων, αλλά και για το σχέδιο που μόλις ανέφερα. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ για την ε, απόφαση να χρησιμοποιούνται περισσότερο επιλεκτικά αλληλευτικά εργαλεία. Και οι μειώσεις 25% όμως να πω ότι ενδέχεται να διαλύσουν τον αλληλευτικό τομέα. Έγραψα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο χρόνια, ιδιαίτερα για το θέμα αυτό, για τη Δυτική Σκοτία και τους παρακάλεσαν να αλλάξουν πορεία, να αλλάξουν κατεύθυνση, διότι αυτές οι μειώσεις του 25% ήταν καταστροφικές για την αλληλεία και οδήγησαν σε ακόμα περισσότερες απορρίψεις. Μου φαίνεται πάντως ότι μπορούμε να βρούμε κάποιο φως στο τέλος του τούνελ εάν προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις. Και ελπίζω να γίνει έτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στίβενσον. Κύριε Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την Επιτροπή για αυτή την παρουσίαση και την εισηγήτρια για τη δουλειά την οποία κάνει πάνω στον κανονισμό. Πολύ θετικό που η Επιτροπή στην πρότασή της όντως καταδεικνύει τα σημεία αυτά στα οποία δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το, ο μηχανισμός και συμφωνώ με πάρα πολλές από τις πτυχές τις οποίες επισημαίνουν. Θα ήθελα επίση να πω ότι βέβαια πρόκειται για ένα νομοθέτημα για να προσαρμόσει το σχέδιο ε, για τα αποθέματα γάδου στην ε, Βαλτική. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο με λίγο βλέποντας ότι θέλετε να έχετε ένα μεικτό ε, σχέδιο για πολλαπλά ήδη το 2014. Αυτό για μένα είναι καινούριο. Νόμιζα ότι θα έφτανε φέτος το Δεκέμβριο. Θέλω να ακούσω αν ισχύει, αν ισχύει τελικά, θα ισχύει για το 2014. Και σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον υπολογισμό των προσπαθειών των αλλιευτικών σκαφών, δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού. Η ανάγκη ευελιξίας σε σχέση με τον κανονισμό για τα αποθέματα γάδου δεν είναι μόνο μια αριθμητική μείωση των ΤΑΚ, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση κατά περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό να τα διαπραγματευτούμε όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και η ανάγκη προσαρμογής του υφιστάμενης νομοθεσία στην συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως, νομίζω ότι είχε η λογική η πρόταση της Επιτροπής, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις υποχρεώσεις μας προς την ε, βιομηχανία της, ε, του τομέα της αλίας. Ας μην κάνουμε μπαλώματα με προσωρινά νομοθετήματα όταν δεν έχουμε παρκή στοιχεία. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία με την ε, εισηγήτρια και τον σκιώδη εισηγητή του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λεβίν. Eh, eh, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την παρουσίασή της. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς μία πρακτική ερώτηση. Εάν εγκρίνουμε την τροποποιημένη πρόταση, τι θα γίνει η πρόταση λησαφωνοποίησης. Θα έχουμε μόνιμα σχεδία διαχείρισης για τον γάδο στη Βόρεια Θάλασσα ή η πρόταση αυτή σημαίνει πως θα ακυρωθεί η άλλη. Και έπειτα, μία ερώτηση σχετικά με το άρθρο 9. Διαβάζοντας το άρθρο 9.2β για την ελαστικότητα, την οποία αναφέρατε, διαβάζω στα αγγλικά. Insufficient information to set attack in accordance with paragraph 1, there might be a reduction of the TAC from the previous year by 25%, or, if scientific advice so recommends, a reduction not exceeding 25% compared to the attack in the previous year, together with other appropriate measures. Förstår jag det här rätt då, att man kan välja mellan att... Εάν κατάλαβα καλά, μπορούμε να επιλέξουμε είτε για μείωση ποσοστού 25% των ΤΑΚ, είτε με κάποιο άλλο ποσοστό. Αλλά τι ποσοστό είναι αυτό, μπορεί να είναι 1% ας πούμε. Πώς θα επηρεάσει αυτό τον γάδο στο Κάτεγατ. Τα αποθέματα γάδου εκεί είναι στα χαμηλότερα επίπεδα που είχαν ποτέ. Μπορείτε να φανταστείτε. Από τη δεκαετία του 1970 μειώνονται τα αποθέματα γάδου εκεί. Από 20.000 τόνους τότε φτάσαμε πέρυσι σε 145 τόνους μόνο. Τα επίπεδα της, μειο... της βιομάζας έχουν μειωθεί δραματικά. Και θα αφήσουμε αυτήν την ε, ελαστικότητα στα κράτη-μέλη να, μειω... να κάνουν μείωση μόνο 1% Δεν γνωρίζω εάν αυτό που φταίει είναι τα ανεπαρκή στοιχεία ή όχι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει η αλία στο κάτεγατ να σταματήσει. Και αυτό, το ότι πρέπει δηλαδή να σταματήσει, είναι βασισμένο σε, επιστημονικές μελέτες ή όχι. Και τέλος. Θα ήθελα να καλωσορίσω αυτά τα καλά νέα από την Νορβηγία για τα αποθέματα γάδου στη Βέργια θάλασσα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Αυξήθηκαν 10 φορές μέσα σε 10 χρόνια. Από 50.000 τόνους σε 2 εκατομμύρια τόνους. Και αυτό είναι 10 φορές πάνω από την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των αποθεμάτων αυτών. Κύριος Βαλέσα, Ο κύριος... Νομίζω ότι ο κύριος Στίβενσον έχει σχετικά σχέδια, αλλά ο κανονισμός του 2008 είναι ένα σχέδιο για την διαχείριση των αποθεμάτων γάδου που δεν γραμμίσει με τρέχουσα πραγματικότητα. Όλοι το γνωρίζουμε και καταδίθηκε στα πλαίσια των συζητήσεων στην Επιτροπή αυτή. Γι' αυτό και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την προτινόμενη αναθεώρηση του σχεδίου και χαιρόμαστε για το ε, τι προτείνει η κυρία Ντότζ. Μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ το περιεχόμενο αυτό που μας παρουσίασε. Το εργαλείο της ευελιξίας είναι εξαιρετικό και εύχομαι κάθε επιτυχία με το σχέδιο αυτό και ελπίζω να έχουμε έξοχη συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Φράγα. Έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση για την Κομισιόν. Εγώ θεωρούσα πάντοτε ότι το πρόγραμμα ανασύστασης του μπακαλιάρου του γάδου ε, ήταν ε, πολύ πιο ήπιο από ό,τι άλλα, όπως αυτό του ερυθρού τόνου. Γιατί η ανασύσταση των αποθεμάτων γάδου που ξεκίνησε ε, από ένα επίπεδο ε, χαμηλότερο του ορίου ε, βιωσιμότητας που δεν είχε και σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση για τον ερυθρό τόνο που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εδώ τώρα τι προτείνουμε, ε, μέγιστη μείωση του 25% ενώ για τον ερυθρό τόνο είχαμε μειώσει στο παρελθόν μέχρι και 40% ενώ η Κομισιόν είχε προτείνει μέχρι και 70% και παραπάνω από 70%. Οπότε δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τη λογική της Κομισιόν. Η Κομισιόν από την άλλη μεριά το 2003 για τη Βόρεια Θάλασσα μια αύξηση του τάκ του μπακαλιάρου. Πώς είναι δυνατόν, μπορεί να το εξηγήσει κανείς αυτό, πώς είναι δυνατόν να προταθεί για τη Βόρεια Θάλασσα ε, αύξηση του τάκ του μπακαλιάρου για αποθέματα που είναι χειρότερα από τα αποθέματα του ερυθρού τόνου και για τον ερυθρό τόνο ε, προτείνονται ακόμα μειώσεις ενώ η Επιστημονική Επιτροπή έχει πει ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν τα τάκα τα 600 τόνους. Γιατί λοιπόν η, ε, αυτή η διαφορά, αυτή η διακριτική μεταχείριση. Ευχαριστώ λόγω στην Κομισιόν να μας διευκρινίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Uh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα μου επιτρέψουν να διευκρινίσω ορισμένα ζητήματα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εισηγήτρια. Σε μια επόμενη συνάντηση μπορούμε να συζητήσουμε λεπτομερώς τις προτάσεις και τις τροπολογίες. Να απαντήσω καταρχήν στην πρώτη ερώτηση. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ε, αν με την ε, πρότασή μας ε, ε, επιταχύνουμε τη διαδικασία. Στο άρθρο 9 η πρότασή μας προβλέπει ότι όλα θα τα προτείνει η Κομισιόν επί τη βάση των επιστημονικών δεδομένων για τα διάφορα αλλιεύματα και τις διάφορες περιοχές. Για... Ε, έχουμε πει ότι θα βασιστούμε στα επιστημονικά δεδομένα. Δεν θα υπάρξει καινούργια διαδικασία συναπόφασης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση, τις πληροφορίες και τα σχόλια που έρχονται από τους επιστήμονες ή κομισιόν, ε, θα υποβάλει τις προτάσεις της. Να επιβεβαιώσω την ερμηνεία της κυρίας Λεβίν. Το 9-2-Β, β δίνει ευελιξία σύμφωνα με την προσέγγιση κατά περίπτωση. Α, θα είναι, ε, η, η μείωση θα είναι από 0 25%. Δεν θα έχουμε πλέον αυτόματες μειώσεις του 25%, αλλά πρώτον θα έχουμε το κριτήριο των επιστημονικών δεδομένων και όταν τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να καθορίσουμε ένα επίπεδο αλλιευμάτων προσπάθειας και δεν έχουμε άλλου τύπου κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, τότε θα προβαίνουμε σε μία μείωση, με ευελιξία όμω, λαμβάνοντα υπόψη όλα τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν για να λυθεί το πρόβλημα του, των συγκεκριμένων αποθεμάτων. Για τη Δυτική Σκοτία και επί τη βάση των καινούργιων επιστημονικών δεδομένων δεν πρόκειται να βρεθούμε ξανά στην κατάσταση που ήμασταν στο παρελθόν δεν θα έχουμε πλέον έλλειψη επιστημονικών δεδομένων. Τα επιστημονικά δεδομένα υπάρχουν πια. Έχουμε μια αναλυτική ε, ε παρουσίαση των δεδομένων και λαμβάνοντας και μπορούμε πλέον να, τα λάβουμε υπόψη για μια, ε, το κατάλληλο επίπεδο μείωσης. Ε, βέβαια, η επιστημονική τα επιστημονικά πορίσματα ζητούν σημαντική μείωση, πλην όμως δεν έχουμε πλέον έλλειψη επιστημονικών δεδομένων. Επί τη βάση των υπαρκτών επιστημονικών δεδομένων πλέον, αναλυτικών μάλιστα, θα προτείνει η Κομισιόν τη μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας. Τώρα, πώς συνδέεται αυτή η πρόταση και η νέα πρόταση. Να σας επαναλαμβάνω ότι αυτή η πρόταση δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Συζητούμε με τους επιστήμονες και θα συνεχίσουμε να συζητούμε και με τους επιστήμονες και με τους φορείς του κλάδου και με τα κρατη έτσι ώστε να ε, καταλήξουμε στο μέλλον σε ένα σχέδιο μικτής αλίας. Γνωρίζουμε, ότι το, για ποιους, γνωρίζουμε ποιες είναι οι αδυναμίες αυτού του σχέδιου Πολλές φορές οι αδυναμίε αυτέ οφείλονται στην κακή εφαρμογή του σχεδίου από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι ε, για τους οποίους το σχέδιο αυτό δεν δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε διάφορα σενάρια και την προσέγγιση, τη μεικτή προσέγγιση προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα του συγκεκριμένου αποθέματος. Δεν νομίζω ότι κάνουμε διάκριση ε, εναντίον του ε, ερθρού τόνου και υπέρ του γάδου. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο καταστάσεις. Ενδεχομένω δεν έχετε τι σωστέ πληροφορίε για τον γάτο στη Βόρεια Θάλασσα. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση εκεί του αποθέματο βελτιώνεται. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα μας επιτρέψει να προτείνουμε αύξηση των, των ποσο, αλλιεύσιμων ποσοτήτων. Αντιθέτως, θα προτείνουμε μείωση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε όμως τις, τα δύο αυτά αλλιεύματα. Θέλουμε με αυτή μας την πρόταση να αποφύγουμε αυτοματοποιημένες μειώσεις. Όταν να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε και άλλα κατάλληλα μέτρα που θα μας επέτρεπαν να βελτιώσουμε την κατάσταση του αποθέματος. Στην πρότασή μας υπογραμμίζουμε την σημασία του να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε, να προσδιορίζουμε και να εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα που θα επιτρέπουν τη χρήση πιο επιλεκτικών εργαλείων για να αποφύγουμε τα υψηλά επίπεδα απορρίψεων που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά θα είναι τα βασικά μέτρα τα οποία θα προσδιορίσουμε και θα εφαρμόσουμε για την βελτίωση των αποθεμάτων σε όλες τις περιοχές που καλύπτονται από το τρέχον ισχύον σχέ, ε, ε, μακροπρόθεσμο σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντότς για να τελειώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Thank you. ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα απαντήσω σε κάποια από αυτά τα οποία θεωρώ σημαντικά. Νομίζω σχεδόν όλοι μας μπορούμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι το σχέδιο ανάκαμψης του γάδου, το οποίο πρωτοτέθηκε σε εφαρμογή το 2008, είχε διάφορα προβλήματα και οι αξιολογήσεις που έγιναν το 2011 έδειξαν πως δεν δουλεύουμε σωστά. Ελπίζω να απαντήσω στην ερώτησή σχετικά με τις δύο εκθέσεις αυτό που έγινε είναι ότι τώρα φτιάξαμε ορισμένες βελτιώσεις με το σχέδιο, σχετικά με το σχέδιο του 2008 και προσπαθούμε να το εναρμονίσουμε με την συνθήκη της Λισαβόνας. Από τη μία, δηλαδή λοιπόν είναι θέμα ουσίας και από την άλλη έκθεση έγινε πολύ πιο τεχνική. Και πιστεύω πως είναι η πιο συνετή λύση να προχωρήσουμε και με τα δύο θέματα παράλληλα. Όσον αφορά με την αυτόματη μείωση 25% στην οποία αναφέρθηκαν οι περισσότεροι από εσά σήμερα. Ε, αυτή η μείωση θα οδηγήσει στο να κλείσουν αλληλευτικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων θα μας βοηθήσει καλύτερα. Δεν θα καθυστερήσει τη διαδικασία. Αντιθέτως, πιστεύω πως θα διευκολύνει αυτήν την πολύ περίπλοκη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Επίσης, Νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι ότι αυτό είναι δεν είναι παρά ένα βήμα προς τα επόμενα αλληλευτικά σχέδια και καλύτερα να γίνουν τώρα παρά αργότερα. Μου λέμε πως το 2014 είναι η καλύτερη εποχή για αυτά τα πολιετή σχέδια και νομίζω πως υπάρχει, θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αν συνεργαστούμε καλά θα μπορέσουμε. Τέλος, να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη μελλοντική μας συνεργασία και παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα χαρώ πολύ να σας συναντήσω προσωπικά και να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τα επιμέρους σχόλια στον τελικό κανονισμό. Ωραία, περνάμε στο σημείο 11. Πρωτοκόλλο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισλαμική Δημοκρατία τη Μαυριτανία σχετικά με τον καθορισμό των αλληλευτικών δυνατοτήτων και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη μεταξύ των δύο πλευρών. Ε, επειδή είμαι εισηγητή, ε, θα ήθελα να ξεχωρίσω το, το ρόλο μου ω πρόεδρο και ω εισηγητή. Γι' αυτό το λόγο δίνω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρο και κατεβαίνω κάτω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα Προεδρεύσω λοιπόν για αυτό το θέμα έτσι ώστε ο εισηγητής ε, να νιώσει πιο άνετα και να μας ε, εκθέσει τα του πρωτοκόλου μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή. Α, στην Επιτροπή πρώτα. Επιτροπή. Obviously. Thank you, Chairman. Ε, <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο ήδη έχει συζητηθεί σε διάφορες ε, περιπτώσεις και ευκαιρίες σε κάποιο βαθμό. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο προκύπτει από μακρές ε, διαπραγματεύσεις και αντίθετα με τους αρχικούς σχεδιασμούς μας κατέληξε σε μια πρόταση να υπάρξει ένα διετές πρωτόκολλο με μια χρηματική συνεισφορά 67 εκατομμυρίων για αλληλευτικές ευκαιρίες και 3 εκατομμύρια για οικονομική στήριξη των ε, Μαυρετανών αλλιέων. Σε σχέση με τις ευκαιρίες αλλιές που προβλέπονται στο πρωτόκολλο, οι κύριες κατηγορίες είναι πελαζικά ε, είδη, ε, οστρακοειδή και τόνος και μια κατηγορία που εισέρχεται κατά περίεργο τρόπο είναι κεφαλόποδα, τα οποία έρχονται με μηδενική ποσότητα που όμως θα αναθεωρηθεί κατόπιν νέων επιστημονικών στοιχείων και νέων αξιολογήσεων που έχουν γίνει από τη Μαυριτανία σε ό,τι αφορά τα διατηθέμενα πλεονάσματα των αλλιευμάτων. Κάτι άλλο το οποίο είναι αξιοσημείωτο σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο είναι μια αλλαγή των τεχνικών συνθήκων. Ήταν ένα θέμα ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς ε, Μαυριτανίας που ήθελαν να έχουν μια σειρά στόχων που θα ε, επιδιωχθούν με αλλαγή των στέχιων αυτών. Καταρχώς στόχος ήταν αύξηση του ελέγχου των ε, αλλιευτικών δραστηριοτήτων, ένας στόχος ο οποίος είναι, ε, το συμμεριζόμαστε απόλυτα. Μετά υπήρχε ένας στόχος διατήρησης των αλλιευμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει λιγότερη επιρροή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βάτο το, το το οποίο οδήγησε στην καθορισμό νέων αλληλευτικών ζωνών. Υπήρξε μια επιπρόσθετη τεχνική συνθήκη η οποία προέκυψε από την ε, επιθυμία της ε, μαυριτανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τον τόπιο πληθυσμό να υποφεληθεί από τις αλληλευτικές δραστηριότητε, ε, ώστε να υπάρχει, ώστε το χρησιμοποιούν σαν τροφή. Είναι πασίγνωστο ότι οι Μαυριτανοί δεν αρέσκονται ιδιαίτερα στο ψάρι και ταυτόχρονα υπάρχει και το, υπάρχει το πρόβλημα σωστής διατροφής του πληθυσμού, του ντόπιου πληθυσμού. Υπήρξε λοιπόν αυτή η κοινοτομία να υπάρξει ε, η συνεισφορά 2% σε είδος να δίνεται και πάλι για την ε, διατροφή του τοπικού πληθυσμού με εξαίρεση των ε, αλλιευτικών ανοιχτής θαλάσσης. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και μια τέταρτη τεχνική προϋπόθεση ήταν να εμπλακεί περισσότερο ντόπιος πληθυσμός στη δραστηριότητα αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία ντόπιων αλλιέων πάνω στα ευρωπαϊκά, στα κοινοτικά σκάφη, τα κοινοτικά αλληλευτικά σκάφη για τις διάφορες αλληλευτικές δραστηριότητε. Αυτές οι τεχνικές προϋποθέσεις, κάποιες εξ αυτών θεωρούμε ότι μπορούν ίσως να αντικατασταθούν από άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι γενικά ευθυγραμμίζονται με τις ε, υποδείξεις που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτού ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση για το πρωτόκολλο αυτό πηγώντας ακριβώς ε, την ε, ίδια κατεύθυνση, ε, συμπεριλάβαμε και τη σχετική σύσταση να αλλάξει η σχετική συνεισφορά του ευρωπαϊκού προπολογισμού και του στόλου, δηλαδή να αυξηθεί η συνεισφορά με το στόλο και ταυτόχρονα κρατήσαμε τη σημείωση ότι όλες αυτές οι αλλαγές των τεχνικών συνθήκων προκαλούν μια κάποια ανασφαλεία για τους στόλους. Άρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προς προσαρμογή. Στη διαπραγμάτευση λοιπόν ζητήσαμε από τη Μαυριτανία να επιτρέψει στον ευρωπαϊκό στόλο να έχει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τους ε, ε, υδρόβιους πόρους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το πελασγικό στόλο, όπου υπήρχε ένα θέμα να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει υπεραλίευση. Προτεραιότητα λοιπόν δίνεται στον ευρωπαϊκό στόλο και ταυτόχρονα τη διασφάλιση ότι αν προκύψουν, αν έρθουν και άλλοι στόλοι θα έρχονται μόνο σε περίπτωση που όντως υπάρχει ε, περίσσια αφού θα έχει καλύψει την ε, ποσόστοσή του Ευρωπαϊκού Στόλου. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην συμφωνία με τη Μαυρετανία. Και επίσης ζητήσαμε η Μαυριτανία να εφαρμόζει τις ίδιες τεχνικές και χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις σε όλους τους τόλους. Όχι εφόσον αποδέχθηκαν δηλαδή να εισάγουν κάποιου όρου. Δηλαδή, ο ευρωπαϊκό στόλο, ο κοινοτικό στόλο έχει προτεραιότητα, αλλά ταυτόχρονα οι τεχνικέ συνθήκε οι οποίε ε, ε, μπαίνουν αυτή τη στιγμή δεν θα οδηγήσει σε μειονεκτική θέση του κοινοτικού στόλου σε σχέση με άλλου στόλου. Λόγω όμως της αβεβαιότητας εισάγαμε και το στοιχείο της ε, καινοτομίας, δηλαδή εξασφαλίσαμε ότι εάν μετά από μια αρχική απόπειρα εργασίας κάτω από τις τεχνικές αυτές συνθήκες, ο ευρωπαϊκός στόλος θεωρήσει ότι δεν είναι επικερδής ε, η όλη επιχείρηση, μπορούμε να καταγγείλουμε το πρωτόκολλο. Υπάρχει δυνατότητα μονομερούς καταγγελίας του πρωτοκόλλου. Υπάρχει δηλαδή μια ρήτρα διασφάλισης που θα μας ε, εξασφαλίσει ότι δεν θα συνεχίζουμε να καταβάλουμε αντιπαροχή εάν δεν εξασφαλίζεται η κερδοφορία σύμφωνα με τους όρους του τρέχοντος πρωτοκόλλου. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την οικονομική υποστήριξη, ξέρετε ότι στο προηγούμενο πρωτόκολλο η δυνατότητα ε, απορρόφησης ε, από πλευρά Μαυρετανία δημιουργήσε πρόβλημα. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζουμε ότι δεν θα καταβληθεί νέα χρηματική βοήθεια εάν προηγουμένω δεν έχουν απορροφηθεί οι πιστώσει οι οποίε έχουν δεσμευθεί για την Μαυρετανία. ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν κονδύλια τα οποία θα παραμένουν χρησιμοποιητά σε λογαριασμού. Αυτή ήταν μια γενική επισκόπηση του νέου πρωτοκόλου. Νομίζουμε ότι εισάγει κάποιες αβεβαιότητες, είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη εισάγει και κάποιες καινοτομίε και επομένως θα πρέπει να εφαρμοστεί για... και θα βέβαια είναι προσδοκιμή από τον κοινοτικό στόλο. Προσκαλούμε το συντομότερο δυνατόν αυτή τη στιγμή σε υιοθετηθεί το πρωτόκολλο να πάει ο στόλος και να δοκιμάσει, να δει τι αποκομίζει, να έρθουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και αν υπάρχει ανάγκη να το συζητήσουμε με τη Μαυριτανία, αν μπορεί να γίνει κάποια προσαρμογή τεχνικών όρων που θέτουν περιορισμούς. Ζητήσαμε από την εταίρο μας, ρωτήσαμε κατά πόσο είναι πρόθυμοι να το κάνουν και είχαμε θετική ένδειξη. Δηλαδή αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει πραγματικά είναι να κρατήσουν την ουσία αυτών των τεχνικών προϋποθέσεων. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες, θα μπορούσε εφόσον βλέπουμε ότι παρεμποδίζουν τις ε, δραστηριότητες, να υπάρξουν, θα μπορούσαν να αποδεχθούν να αλλάξουν κάποιες συνθήκες, όπως για παράδειγμα την αλληλευτική προσπάθεια, την απόδοση αλλά αλληλευτική προσπάθεια κλπ. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό είναι να δούμε ότι μέσω αυτού του πρωτοκόλου μπορέσαμε να καθοδηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο προς την επιθυμητή κατεύθυνση τη Μαυριτανία, πράγματα που τον επιθυμητό και από το Κοινοβούλιο αυτό, και σε ό,τι αφορά την διατήρηση των αλλιευμάτων και για την επανεξορρόπηση των χρηματοοικονομικών συνθήκων και μπορέσαμε να εξάγουμε τις συνθήκες αυτέ και προς ε, άλλα ε, μέρη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εμεί θέτουμε του κανόνε. και στόλοι που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή της Μαυριτανίας πρέπει να υιοθετήσουν τους κανόνες αυτούς. Εάν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσει, ευχαρίστω να απαντήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντεπιπέρ. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεπιπέρ. Πράγματι έχουμε μιλήσει πολύ για αυτό το ζήτημα για μήνες Οπότε δεν θα μακρηγορήσω. Ε, Επίση έχουμε μιλήσει πιο πολύ για το τι ήθελε η Μαυριτανία και λιγότερο για το τι θέλουμε εμείς. Όμως αυτή η συμφωνία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον. Καταρχήν ότι ε, η Κομισιόν τη διαπραγματεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Κοινοβούλιο και τον κλάδο. Και δεύτερον, ότι ο κλάδος, ο κλάδος δεν τη θέλει αυτή τη συμφωνία και το έχει πει και προφορικά και γραπτός. Την περασμένη εβδομάδα πριν από μερικές μέρες το είπανε και προφορικά στην Επίτροπο. Όλα αυτά θα ήταν, έπρεπε να είναι αρκετά για να αναθεωρήσει τη στάση της Κομισιόν και να ε, αποφασίσει να μην προχωρήσει με την ε, επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Όλα αυτά είναι σαφή. Ε, να σας αναλύσω τι, ποια είναι η άποψη του κλάδου. Έχουμε μια συμφωνία που υπογράφηκε για δύο χρόνια, μετά από μια διαπραγμάτευση περίπου δύο ετών. Βλέπουμε ποιοι είναι οι ρυθμοί. Ε, δεν μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική βέβαια αυτή η συμφωνία. Κοστίζει 70 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πέραν του, των ποσών που πληρώνονται για τις άδειε. Ένα νέο κόστος το οποίο είναι τριπλάσιο σε σχέση με το τι κόστιζε η άδεια μέχρι τώρα. Επίση έχουμε πρόβλημα και με τις αληφτικές περιοχές. Νομίζω ότι ο κλάδος το είχε πει πολύ καθαρά να μην αλλάξουν οι περιοχές γιατί αλλιώς ε, τροποποιεί το πάρα πολύ και μειωνόταν η αποδετικότητα. Ε, και, και ο καθεσμός, το, ε, ο ημείος των 6 μιλίων και οι ίδιες συντεταγμένες των περιοχών που προβλέπονται είναι τέτοιες πλέον με την καινούργια συμφωνία που δεν είναι βιώσιμη. Ούτε τα ε, συγγνώμη, τα αλληλευτικά ε, είδη δεν κινδυνεύουν, ποτέ δεν ελέγχθηκε κάτι τέτοιο, παρόλα αυτά εφαρμόζονται τάκ, ε, που επιπλέον θα είναι και πολύ πιο περίπλοκο να εφαρμοστούν. Θα Ε, Πιστεύω ο κλάδος ότι ε, συνεχώς ε, θα του επιβάλλονται κυρώσεις και, σίγουρα η κατάσταση δεν θα είναι πολύ σαφής. Μετά, τα παραλιεύματα μειώνονται πάρα πολύ. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά σημαντική οικονομική ζημία για τον κλάδο. Αν σε αυτή την κατάσταση προσθέσουμε το μονοπόλιο των του, καυσίμου, οι υποχρεώσεις φόρτωσης εκφόρτωσης ε, και, διάφοροι άλλοι, και διάφορους άλλους περιορισμούς, η κατάσταση χειροτεύει ακόμα περισσότερο. Κανένα δεν αμφισβητεί λοιπόν ότι όλα αυτά είναι αρνητικά για τον κλάδο. Λέγεται ότι υπάρχει και κάποιο, υπάρχουν και κάποια θετικά. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω. Ε, δεν επικρίνω τους διαπραγματευτές, έχει και θετικά σημεία η συμφωνία, αλλά δεν είναι αρκετά. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον ελεκτικό στόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να δούμε στην πράξη τι θα σημαίνει αυτό, ότι ο δικό μας στόλος θα έχει προτεραιότητα. Ε, θα το δούμε στην πράξη αυτό. Μετά, η ρήτρα διαφύλαξη, η οποία μα επιτρέπει να, μας επιτρέπει να μην πληρώσουμε. Εδώ είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Το πρωτόκολλο λέει ότι ε, θα πρέπει οι η πληρωμή να γίνει τρεις μήνες μετά την επικύρωση. Όλα αυτά λοιπόν τα 70 ε, εκατομμύρια θα πρέπει να πληρωθούν σε τρεις μήνες. Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη εγγύηση είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα αν οι συνθήκες ε, ε δεν είναι αυτές που περιμέναμε ότι δηλαδή τα αλλιεύματα δεν είναι τόσα όσα προβλέπονται ε, τότε μπορούμε να ε, πληρώσουμε μικρότερες ποσότητες. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε πώς αυτό θα εφαρμοζόταν. Απ' την άλλη μεριά, αν μέσα στους τέσσερις μήνες που μας δίνονται πράγματι κοινοποιήσουμε μια τέτοια ε, υποαπορρόφηση, μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε. Γιατί να επαναδιαπραγματευτούμε, γιατί να περιμένουμε λέω. Αφού ο κλάδο μα ζητάει ήδη να επαναδιαπραγματευτούμε, γιατί να περιμένουμε 4-5 μήνε και να επενδύσουμε 70 εκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι θα γίνουν όταν θέλουμε έτσι κι αλλιώ να επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία. Αν υπάρχει πολιτική βούληση να επαναδιαπραγματευτούμε, γιατί να μην το κάνουμε ήδη ε, πριν δώσουμε και τα χρήματα, αντί να το κάνουμε αργότερα. Ε, είναι εύκολη απάντηση αν υπάρχει πολιτική βούληση. Μας λένε, ήταν η πιο καλή ε, συμφωνία μπορούσαμε να πετύχουμε. Παρόλα αυτά, και δεν θα μπω σε θέματα τύπου κεφαλόποδα κλπ. Το αν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιστημονικές μελέτες για το κατά πόσον το είδος αυτό κινδυνεύει όχι. Εν πάση περιπτώσει δεν θα μπω σε αυτό το θέμα. Γιατί και εκεί το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Ήδη όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας ανέφερα είναι αρκετά σημαντικά και αρνητικά. Η Κομισιόν λέει ότι είναι διαθέσιμη να συζητήσουμε, είναι πρόθυμη ε, και το καταλαβαίνω αυτό γιατί η Κομισιόν έχει αντιληφθεί πως υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία πάρα πολύ αρνητικά πολύ βλαβερά, ακόμα και στις, ε, στις, ε, στους τεχνικούς όρους. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό τώρα όμως. Γιατί να μην ξεκινήσουμε την επαναδιαπραγμάτευση τώρα. Θα ήθελα να μου πει ποια είναι η πρόθεση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις ε, προθεσμίες, τους τρόπους πληρωμής, τη δυνατότητα να αποφύγουμε την πληρωμή κλπ. Και επίσης ε, τι πιστεύει η Κομισιόν για όλα αυτά που έχει ακούσει από την μεγάλη πλειοψηφία του ίδιου του κλάδου. Είδα και την ίδια την επιστολή που έστειλε, ε, έστειλε ο κλάδος στην Επίτροπο. Για, την, ε, για το γεγονός ότι ο κλάδος θεωρεί πως η συμφωνία αυτή οικονομικά δεν είναι προσοδοφόρα. Αυτό που θέλαμε είναι μια... Αυτό που θέλουμε είναι μια συμφωνία καλύτερα από αυτή που έχει αυτή τη στιγμή επικυρώσει η Κομισιόν. Έχει υπογράψει η Κομισιόν, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε συνάλφοι θέλουν το λόγο. Κύριος Βαλέσα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα πολύ σύντομο ερώτημα, το οποίο εξακολουθεί να μου τριβελεί στο μυαλό. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει μια συμφωνία με την Βρετανία και να ενθαρρύνει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να την ε, υιοθετήσει τη συμφωνία αυτή, με την σαφή άρνηση όμως ε, της Μαυριτανίας ό,τι αφορά τα πελαγικά είδη. Θέτω και πάλι το ερώτημα αυτό, γιατί δεν μπορώ να το κατανοήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Λαβάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Καμπριέλ, για την παρουσίασή σου. Δεν συμφωνώ όμω καθόλου μαζί σου ότι πρέπει να αρχίσουμε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής. Νομίζω ότι το πρωτόκολλο εν πολλής βασίζεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σέβεται όλα όσα έχουμε συμπεριλάβει στο ψήφισμα εκείνο και υπάρχουν σαφέστατες αρχές οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παραδιαπραγμάτευση. Έχουμε δηλώσει ότι πρέπει να σεβαστούμε τις αρχές αυτές. Υπάρχουν ε, σχετικές, ε, σχετική προβληματική σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και δεν θα πρέπει να υπάρχει περιελίευση και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο πρωτόκολλο αυτό. Μια σαφέστατη αρχή είναι ο σεβασμό και το ότι δεν θα πρέπει να έρθουμε σε ανταγωνιστική θέση με τους ντόπιου αλείς και να ε, διακινδυνεύουμε βέβαια την επιστημιστική ασφάλεια των χωρών αυτών. Και στα θέματα των κεφαλόπεδων υπήρξε σαφέστατο αίτημα από τον κλάδο της μικρής κλίμακας ε, αλληλείας στη Μαυριτανία. Υπάρχει αίτημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που διατείνονται ότι τελικά ο κοινοτικός ε, ε, στόλος α, τους ανταγωνίζεται. Ζητούσαν πάντα ε, να εξαιρεθεί το χταπόδι και όντως έχει γίνει στο πρωτόκολλο αυτό. Ε, έχουν τα μεγάλα σκάφη ανταγωνίζονταν με την ε, εξωτερικού στόλου στην Ιαπωνία για παράδειγμα για την αλίευση χταποδιού και υπάρχουν πλέον ε, αλλιεύματα τα οποία απολούνται στην ίδια τη που προέρχονται από κοινοτικό στόλο σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι μπορούν να το διαθέσουν οι ντόπιοι αλληλείς. Αυτό δεν μπορούμε να το πάμε να διαπραγματευτούμε. Αυτό είναι θέμα αρχή και το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη. Πρέπει να σεβόμαστε συγγνώμη, τον ντόπιο πληθυσμό. Και βέβαια πρέπει να εξασφαλιστεί η ψηφιστική ασφάλεια, γιατί είναι πολύ ισχυρότατη αρχή και θέλω να ευστήσω, στην, ευστήσω την προσοχή σας ότι υπήρξε στην Μαυριτανία, στην Αξότ, μια συζήτηση, ένα φόρουμ, όπου η συζήτηση των πολιτών και ο κλάδος της Αλίας ήρθαν σε επαφή. Ε, συζήτησαν 14 και 15 ε, Οκτωβρίου, μόλις πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή και εξέδωσαν την δήλωση αυτή και συστάσεις όπου εν πολλής υποστηρίζουν το τρέχον πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα σημεία του. Για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό σημάδι, σημαντική ένδειξη ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με τις ε, ε πολιτικές, ε, εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο κλάδος ε, της αλίας, των αλλιέων στη Μαυριτανία ε, εκτιμά και αποδέχεται το πρωτόκολλο αυτό, για μένα είναι πολύ θετικό και πρέπει να το αποδεχθούμε με χαρά. Δεν βλέπω λοιπόν τι υποτίθεται ότι πρέπει να παραδιαπραγματευτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πρωτόκολλο καταφέρνει ουσιαστικά να συμπεριλάβει την αρχή της μη διάκρισης όλων των αλλοδαπών στόλων, καταδεικνύει ακριβώς ότι επιτύχαμε αυτό που θέλαμε και ζητούσαμε στο ψήφισμα σε ό,τι αφορά την μελλοντική συμφωνία Λίας με τη Βρετανία. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θα έχει την ηγεσία σε έναν αγώνα προς την κορυφή, όχι προς τα κάτω. Να πούμε δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι στόλοι μπορούν να αλλιεύουν μέσα σε τρία μίλια από την παράκτια περιοχή της Μαυριτανίας και επομένως να αφήσουμε όλους τους άλλους στόλους να ανταγωνίζονται με τον τόπιο αλλιευτικό στόλο της Μαυριτανίας και επομένω γιατί να μην το κάνουμε και εμεί. Τώρα, αντίθετα, πλέον η ίδια η Μαυριτανία δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν άλλον στόλο να πλησιάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό την παράκτια περιοχή τη. Και δεν βλέπω πώ μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε τι αρχέ αυτέ. Είναι αρχέ τι οποίε έχουμε όλοι προσυπογράψει. Και εάν αυτό δεν καταστήσει επικερδή τον κλάδο, εάν ο κλάδος χρειάζεται να, να παραβιάσει αρχές δικαιοσύνης και περιβαλλοντικές αρχές, τότε λοιπόν πάρα πολύ ο κλάδος. Αυτός καθ' αυτός είναι περιττός και θα πρέπει να δει πώς θα εξαλείψει σταδιακά τι αδειότητέ του. Γιατί χορηγούμε 70 εκατομμύρια ευρώ κατέτος για να τους βοηθήσουμε να έχουν δηλαδή αλληλευτικέ ευκαιρίες ω αναπτυσσόμενη χώρα. Δεν μπορούν να παραπονιόνται, λοιπόν. Ευχαριστούμε Ισαβέλα. Γιάννα Μιράντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δική μου γνώμη είναι λίγο διαφορετική. Ο αποκλεισμό του, ε, του στόλου των κεφαλοπόδων είναι πραγματικά ντροπή. Ε, πέντε ε, κοινοβουλευτικά ερωτήματα εστέθησαν στην κυρία Επίτροπο για το θέμα των κεφαλοπόδων και το στόλο της Γαλλικίας. Πάνω από 400 άτομα αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν τις ε, ενισχύσεις τις οποίες έχει εγκρίνει η ε, κυβέρνηση και εξαρτώνται από του, τα κεφαλόποδα και προφανώς επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτή την ε, απόφαση και δεν έχουν αλλακτικές λύσεις. Είναι, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος στόλος να χρησιμεύσει σε κάτι άλλο. Στις, 11, στις 5 Οκτωβρίου η Κομισιόν στην απάντησή της λέει ότι είναι δυνατόν το πρωτόκολλο να συμπεριλάβει ρήτρα αναθεώρησης για να ζητήσουμε αλλιευτικές δυνατότητες σε περίπτωση ε, που γίνει ανασύσταση των ε, αλλιευμάτων. Πόσο είναι δυνατόν με βάση τις επιστημονικές έρευνες του Ισπανικού Κοινογραφικού Ινστιτούτου να ενημερώνουμε με σαφή στοιχεία την Κομισιόν ότι, ε, ότι δεν γίνεται υπεραλίευση των κεφαλοπόδων ε, πώς είναι να τον λέω, αυτά τα στοιχεία να μην έχουν ληφθεί υπόψη έγκαιρα. Επίση, αυτοί οι 400 άνθρωποι αλλοί, οι οποίοι δεν λαμβάνουν ενισχύσει, που βλέπουν γκρίζο το μέλλον τους, ε, βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη επαρκώς τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία δώσαμε εμεί στην Κομισιόν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη σήμερα τουλάχιστον αυτές οι επιστημονικές εκθέσεις στη ρήτρα αναθεώρησης. Ο Ολλανδικός τύπος του τελευταίου μήνες λέει ότι ο Ολλανδικός στόλος δεν θα αγοράσει ε, τις ε, ε, άδειε που του αναλογεί γιατί ο κλάδος αντιτίθεται. Είναι δυνατόν να επαναδιαπραγματευτούμε την συμφωνία αυτή. Thank you very much, Mr. Πολύ, ο κύριος Eh, Ο κύριος Σάντσες. Ο πρόεδρος μου δίνει το λόγο, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον παραχωρήσω βέβαια. Η πρώτη συμφωνία με την Μαυριτανία υπογράφηκε το 1987. Είναι το η πιο σημαντική ελευτική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα ζητήματα που γνωρίζω είναι ότι ένα από τα πρωτόκολλα που υπογράφηκαν φέτο τον Ιούνιο έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, αλλά το, το πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία μόνο δύο. Ο κλάδος όμω περιμένει να έχει πιο πλατή ορίζοντα. Για να προγραμματίσει δραστηριότητε του δύο χρόνια δεν είναι αρκετά. Είναι πολύ περιορισμένο, περιορισμένη η διάρκεια αυτής της συμφωνίας. Συμφωνούμε ότι οι σχέσεις με τρίτες χώρες αλληλευτικές σχέσεις με τρίτες χώρες θα πρέπει να μπαίνουν στο πλαίσιο της ε, βιώσιμης ε, ε, διατήρησης των αλευτικών πόρων. Όμως η συμφωνία αυτή δεν νομίζω ότι σέβεται αυτούς τους στόχους. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Δεν γνωρίζω των αλλιών της Μαυριτανίας θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο να μπορούσαν τουλάχιστον να εκφραστούν ε, δημοκρατικά και ελεύθερα. Αλλά γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η γνώμη του κλάδου. Στην ε, Ισπανία, στην περιοχή μου. Και δεν μιλώ για κάποιους μεγαλοαλείς, μικρό, μιλώ για επαγγελματίες ε, ε, ε μικρούς, 400 συγκεκριμένα άτομα που ζουν από την αλία στην περιοχή μου, από την αλία κεφαλόποδων. Ε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλίευαν κεφαλόποδα και όχι μόνο ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες χώρες που αλίευουν κεφαλόποδα στη Μαυριτανία και ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν για ποιο λόγο δεχτήκαμε τον αποκλεισμό των κεφαλόποδων από το πρωτόκολλο. Μου έχει πει η Κομισιόν ότι έλαβε υπόψη της τα, τα πιο επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα. Όταν όμως μπήκα στην σελίδα στην οποία ακριβώς καταγράφονται τα επιστημονικά δεδομένα, <laughs> αυτά τα φοβερά επιστημονικά δεδομένα ε, στα οποία βασίστηκε η ε, Κομισιόν ε, χρονολογούνται από το 2009. Το 2008 μάλιστα υπήρχε μια μικρή μείωση, αλλά το 2009 υπήρξε αύξηση και δεν λύθηκαν υπόψη τα επόμενα χρόνια, 2010, 2011 και φέτος, που δείχνουν ότι τα λιεύματα βρίσκονται σε σταθερότητα και μάλιστα αυξάνονται, τα αποθέματα αυξάνονται κιόλας. Συνεπώς, τα επιστημονικά δεδομένα ε, δεν δικαιολογούν ε, την ε, απαγόρευση της αλληλευτικής δραστηριότητα. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι κάτι πρέπει να γίνει, αυτό θα ήταν μια μείωση, όχι όμως και πλήρης απαγόρευση της αλληλεύσης κεφαλοπόδων. Η ΔΕ Κομισιόν δεν έχει ως ρόλο να προστατεύει τα συμφέροντα των αλλιών της Μαυριτανίας. Μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι, οι Λίβοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Κορεάτες ψαρεύουν εκεί κεφαλόποδα. Και η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η ίδια η Μαυριτανία ε, έχει ε, ε, με τη δική της σημαία σκάφη τα οποία στην πραγματικότητα ανήκουν σε άλλους τόλους τρίτων χωρών. Συνεπώς δεν ξέρουμε ποιανού ακριβώς συμφέροντα ε, είναι αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι συμφέροντα των ε, αλλιών της Μαυριτανίας. Εν πάση περιπτώσει, ε, οι αποφάσεις της Κομισιόν θα πρέπει να είναι λογικές κατά τη στιγμή της αξιολόγησης των πόρων. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 70 εκατομμύρια ευρώ στη Μαυριτανία για την αλία στα ύδατά τη, Όταν ήρθε εδώ η επίτροπο, μα ενημέρωσε για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσει, εμεί είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνουν δεκτές υπερβολικέ οικονομικέ απαιτήσει από πλευρά τη Μαυριτανία. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ δυνατότητε, αληφτικές δυνατότητε που μα δίδονται. Και τι έγινε τελικά. Διατηρείται η, ε, η, η χρηματική αντιπαροχή Ε, αυξάνονται μέχρι τριπλασιάζονται ε, οι τιμές των αδειών και ταυτόχρονα μειώνονται οι αλευτικές δυνατότητε που μας παραχωρούνται. Γίνονται πολλές μειώσεις, για παράδειγμα, στις γαρίδες μέχρι και 25% για αλλιεύματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ε, έχουμε όρους οι οποίοι είναι υπερβολικοί. Ε, διπλός έλεγχος από δορυφόρο για παράδειγμα. Μονοπόλιο ε, στον εφαδιασμό με καύσιμα. Οι αλληλείς μας θα, παίρνουν, θα αγοράζουν καύσιμα πιο ακριβά. 60 ώρες στη θάλασσα ο καθένας τουλάχιστον, ε, όλοι αυτοί οι όροι δεν βοηθούν, δεν προωθούν την ιδέα της ε, ε υγιούς Όλα αυτά είναι στοιχεία πολύ σοβαρά που καθιστούν ε, πολύ προβληματική την τόσο σημαντική αυτή η αλευτική συμφωνία. Θα πρέπει να την αναθεωρήσουμε. Θα ήθελα η Κομισιόν να αναθεωρήσει τη συμφωνία αυτή και να καλέσει τι μαυριτανικέ αρχέ επίση να αναθεωρήσουν το πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Τώρα ο λόγο είναι στην κυρία Πατράου Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τον γενναίο τρόπο με τον οποίο μας, και αντικειμενικό τρόπο με τον οποίο μας παρουσίασε αυτό το σχέδιο συμφωνίας. Ε, πάντοτε είμαστε σκεπτικοί έναντι τέτοιου είδους συμφωνιών. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, συνεπώς ε, δεν εκπλήσει που η άποψή μας είναι επικριτική και για αυτή. Είναι η χειρότερη από συμφωνίες που μας έχει παρουσιάσει η Κομισιόν. Συστηματικά, σε περιπτώσεις διαπραγματεύσεων, σε τέτοιους περιπτώσεις, βλέπουμε μια μείωση των ελευτικών δυνατοτήτων και αύξηση του τιμήματος που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη του αλευτικού τομέα των τρίτων χωρών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα για να δίνουμε χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Γιατί αλλιώς Ας μας ονομάσουν κάτι άλλο. Ας το ονομάσουμε μάλλον το κείμενο κάτι άλλο. Όχι όμως αλληλευτική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα ποσό 70 εκατομμυρίων ευρώ να φεύγουν από τα οθυσαυροφυλάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντιστάθμισμα μια, ε, ένα τίποτα, ένα, μια, μια χούφτα που είναι άδεια. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μια τέτοια συμφωνία, με μια τέτοια αλληλευτική συμφωνία. Γνωρίζουμε την σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση την οποία διανύουμε. Γνωρίζουμε ότι πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, απασχολείται με την ε, μείωση των δαπανών χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών. Πώς είναι δυνατόν, με δεδομένη αυτή την κατάσταση, να υπογράφουμε μια τέτοια συμφωνία που μειώνει τις αλλιευτικέ ε, δυνατότητες που μας δίνονται στο μηδέν σχεδόν. Εκτός η γαρίδα, εκτός τα κεφαλόποδα, συγγνώμη, εκτός ο αστακός, εκτός τα κεφαλόποδα, ε, τι θα ψαρεύουμε, νερό. Ίσως κάποιοι να πιστεύουν ότι αξίζει να ψαρεύουμε νερό. Όμως αυτή η συμφωνία είναι αλλιευτική συμφωνία. Βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντική μείωση των ελευτικών δυνατοτήτων, πλήρης αποκλεισμό κάποιων ειδών από τη συμφωνία, που είναι ε, για, για ιδιαίτερα, τα οποία, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ευρωπαϊκούς αλευτικούς στόλους, βλέπουμε επιδίνωση, γενικότερη επιδίνωση των όρων και του κόστους για τους πλειοκτήτες. Τα ανέφερε ο εισηγητής, πολύ σωστά. Οπότε από οικονομικής πλευράς δεν είναι πλέον βιώσιμο, δεν είναι πλέον ρεαλιστικό να συνεχίσουν να αλλιεύουν στη Μαυριτανία. Για να συνεχίσει ο στόλος μας να αλλιεύει και να μην πρέπει να ψαρεύει όλο και περισσότερο, θα πρέπει τα αλλιεύματα να έχουν συγκεκριμένη ψηλή αξία. Δηλαδή τα αλλιεύματα τα οποία ψαρεύουμε να είναι τέτοια αξία έτσι ώστε να μπορούν, μπορεί να επιβιώσει ο στόλος μας. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να ψαρεύει όλο και περισσότερο από αλλιεύματα χαμηλότερης αξίας. Δεν καταλαβαίνω πώς η Κομισιόν μας υποβάλλει τέτοιου είδου συμφωνία προς ψήφιση. Από αυτή τη συμφωνία δεν είναι δυνατόν να προκύψουν ε, προσοδοφόρες, ε, κερδοφόρες δραστηριότητε. η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, υποστηρίξει τον αλληλευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα ε, να βοηθήσει και τις τρίτες χώρες. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στην βιωσιμότητα των πόρων, ε, των ελευτικών πόρων στη συγκεκριμένη περίπτωση, να δίνουμε παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε και αφελείς ή τυφλοί. Και δεν σημαίνει ότι θα είμαστε οι μόνοι εμείς σε όλο τον κόσμο που θα δίνει το παράδειγμα. σε σημείο ώστε να πληρώνουμε χωρίς να παίρνουμε αντιστάθμισμα. Χωρίς αντίτιμο. Γιατί οι συμφωνίες με όλες τις άλλες χώρες είναι τελείως διαφορετικές. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να είναι ίδια με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά θα πρέπει να πείσουμε, να είμαστε διδακτικοί, έτσι ώστε να πείσουμε τις, τους εταίρους μας, έτσι ώστε οι συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε μαζί τους να είναι ε, κερδοφόρες και για μας. Η Λιβύα, η, η, Ιαπωνία, η Κίνα, η, Νέα, η Νότιος Κορέα δεν βρίσκονται εκεί για να χρηματοδοτήσουν τον ελευτικό τομέα της Μαυριτανίας. Βρίσκονται εκεί για να βγάλουμε κέρδος. Και εμείς πιστεύουμε ότι αν είναι δυνατόν θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε αυτή τη συμφωνία. Και νομίζω ότι είναι δυνατόν. Και αυτή η επαναδιαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνει τώρα. Δεν έχει νόημα να πληρώσουμε πρώτα και μετά να την καταγγείλουμε. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πέραν του οικονομικού, ε, θα είχαμε και θέμα απώλειας διαπραγματευτικής ισχύω. Και εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάμε ότι ε, το Κοινοβούλιο έχει αυξημένη ευθύνη. Ε, αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ένα μοντέλο και για επόμενες συμφωνίε που θα έρθουν προ ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, είμαι υπέρ τη άμεσης επαναδιαπραγμάτευσης αυτής της συμφωνία. Δεν θέλω να τη δεχτούμε έτσι όπως είναι διατυπωμένη αυτή τη στιγμή. Ε, Κυρία Φράγα. Ε, η ουσία κάθε αρχική συμφωνία είναι το εμπορικό κομμάτι. Σε αυτή την περίπτωση η εμπορική συμφωνία από την αρχή των διαπραγματεύσεων ε, βρήκε αντιμέτωπο όλο τον κλάδο. Και από τους τρεις τόλους ε, και το στόλο των ε, κεφαλόποδων και τον στόλο των ε, παραγαδιάρικων και το στόλο των λευτικών σκαφών Αστακού. Στην τελευταία συνάντηση που έγινε, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, και οι εθνικές αρχές και οι πρόσωποι του κλάδου είπαν στην Κομισιόν να μην υπογράψει αυτή τη συμφωνία και τελικά την υπέγραψε. Αντίθετα με τη γνώμη όλων των, των ενδιαφερομένων και των εθνικών αρχών και τοπικών αρχών και των εκπροσώπων του κλάδου. Πέραν αυτού, αυτό που είδαμε ήταν μια απουσία διαφάνειας κατά τη διαπραγμάτευση, γιατί από το Φλεβάρι, και εγώ ήμουν παρούσα στο ΡΑΚ των μεγάλων αποστάσεων που έγινε στις Βρυξέλλες το Φλεβάρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το ΡΑΚ για όλα τα σημεία της διαπραγμάτευσης ε, με λεπτομέρεια. Όταν όμως ήρθε εδώ η Επίτροπος και την ρωτήσαμε ε, τι είναι ανοιχτό και τι είναι κλειστό, μας είχε πει ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στη διαπραγμάτευση, ενώ στην πραγματικότητα ε, είχε επέλθει συμφωνία σχεδόν σε όλα. Μόνο το οικονομικό ήταν ανοιχτό τότε. Είναι λοιπόν μια συμφωνία με την οποία διαφωνούν και οι, οι τρεις τύποι ε, αλληλευτικών στόλων. Ε, ο στόλος για τα κεφαλόποδα προφανώς ε, δεν έχει καμία ποσόστοση. Ε, τα τεχνικά μέτρα από την άλλη μεριά δημιουργούν σημαντικά προβλήματα με τα παραγαδιάρικα. Με το στόλο αλληλείας αστακού επίσης γιατί μειώνται πολύ ποσοστό τους. Τι γίνεται με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα, ε, μάλλον, ε, το ψήφισμα ζητούσε ε, να ληφθούν υπόψη τα πιο σύγχρονα, ε, τα πιο επίκαιρα στοιχεία. Και όμως η Κομισιόν βασίστηκε στα επιστημονικά στοιχεία του 2008. Και είπε κεφαλόποδα μηδέν γιατί η κατάσταση στα κεφαλόποδα ήταν πολύ άσχημη. Τώρα μας, μας τα αλλάζουν και λένε ότι δεν συμπεριλήφθησαν τα κεφαλόποδα επειδή δεν το ήθελαν οι Μαυριτανοί. Όχι, τότε μας έλεγαν άλλα πράγματα. Ότι τα αποθέματα κεφαλόποδων κινδύνευαν. Όμως τα επιστημονικά στοιχεία ήταν διαφορετικά και το Κενογραφικό ε, Ινστιτούτο της Ισπανίας το απέδειξε. Τώρα, στο ψήφισμα επίσης είχε ζητηθεί η τα τεχνικά μέτρα να είναι αντίστοιχα των αλληλευτικών δυνατοτήτων. Γιατί σε τι χρησιμεύουν οι αλληλευτικές δυνατότητες αν με βάση τα τεχνικά μέτρα δεν μπορεί να γίνει αλλίευση. Και εδώ βέβαια έχουμε ε, μια κατάσταση πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Τα τεχνικά μέτρα δεν ευθυγραμμίστηκαν με τις αλληλευτικές δυνατότητες. Τώρα, η Κομισιόν λέει ότι στη, στη Μικτή Επιτροπή μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Όμως το Κοινοβούλιο δεν ζητά αυτό το πράγμα. Το Κοινοβούλιο λέει ότι τα τεχνικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαπραγμάτευση και στη συμφωνία πλαίσιο. Όχι να μην καθορίζονται με βάση τις ε, Μικτές Επιτροπές. Ε, γιατί οι Μικτές Επιτροπές δεν είναι γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που λέει η Κομισιόν δεν είναι η σωστή διαδικασία. Και είδαμε τι έγινε και με την προηγούμενη συμφωνία του Μαρόκου. Και η Κομισιόν είχε πει ότι η ε, Μικτή Επιτροπή μπορούσε να λύσει το πρόβλημα ε, του, ε, ε, του, της αλίας με, με λαμπάρα, ε, αλλά το Μαρόκο είπε εφόσον το έχουμε διαπραγματευτεί δεν πρόκειται να το ξαναδιαπραγματευτούμε. Η συμφωνία με τη Μαυριτανία αντι, ε, αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του συνολικού ποσού που έχει προβλεφθεί στον προπολογισμό για, το, για τις αλληλευτικές συμφωνίες. Θα ήθελα λοιπόν να την επαναδιαπραγματευτούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φράγκα. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γιατί με κοιτούν. <clears throat> Um, Κάποια σημεία που θέλω να διευκρινίσω. Το πρώτο, στη Μαυριτανία. Οι στόλοι μα είπαν δύο πράγματα. Αφενό μας είπαν ότι δεν μα άρεσαν αυτέ τι τεχνικές προϋποθέσεις, αλλά το δεύτερο είναι ότι θέλουμε οπωσδήποτε τη συμφωνία αυτή. Το μήνυμα λοιπόν ήταν ανάμεικτο. Δεν ήταν δηλαδή τα σηκώνουμε και φεύγουμε. Ήταν ε, πολύ πιο λεπτές οι αποχρώσεις. Άρα το ερώτημα ήταν τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Δοκιμάζουμε δεδομένου στις ε, του καινοτόμου στοιχείου αυτών των νέων ε, συνθήκων, να προσκαλέσουμε τους τόλους να δοκιμάσουν και να δούμε τι θα γίνει ή να την άξουμε τη συμφωνία στον αέρα. Οπότε να είμαστε σίγουροι ότι αποκλείεται να υπάρξει οποιαδήποτε αλίευση στον επόμενο χρόνο. Αυτό ήταν το ερώτημα. Το ξέρω ότι υπήρξαν πιο απλές λύσεις, γιατί δεν πάτε στα αεροπλάνο, ελάτε, πιέντε, πιέστε τους, πείστε τους και μετά γυρίστε για να, και να τα έχουμε όλα έτοιμα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι άσπρο μαύρο. Αυτή ήταν μια πρώτη παρατήρηση. Υπήρξαν πάρα πολλές αλλαγές τεχνικές ε, προϋποθέσεις. Υπήρχε μια αύξηση της συνεισφοράς του στόλου. αυτό δεν είναι το κύριο εμπόδιο για τον στόλο. Έχουμε λάβει υπόψη τις ε, οικονομικές συνθήκες και έχουμε λάβει υπόψη την αξία, αν θέλετε, των ε, ηχθείων που έχουν ανέβει τώρα που το υπολογίζουμε σε σχέση με το βάρο και δει σε σχέση με προηγούμενα πρωτόκολλα ή του 87. Καταλαβαίνουμε ότι έχει ανέβει η τιμή των ε, σαριών στην αγορά και προφανώ αυτό το ξέρουν και οι Μαυριτανοί και ήταν λογική η παρατήρησή του και αξίζει να γίνει αποδεκτή. Υπάρχουν λοιπόν αλλαγέ στι τεχνικέ ε, συνθήκε που είναι διαφορετικές ανάλογα με τα τμήματα της αγοράς. Ας πάρουμε τα απελαγικά είδη. Ε, ε, εκπλήσωμαι που δεν βλέπετε να υπάρχει τίποτα σε αντιστάθισμα. Η ποσότητα των πελαγικών ε, αυξάνεται πάρα πολύ. Έχουμε 3.000 τόνους πελαγικών αλλιευμάτων με τη συμφωνία αυτή. Και έχουμε εμεί την προτεραιότητα στα αποθέματα αυτά. Εκπλήτωμαι. Πώς λέτε ότι δεν έχουμε τίποτα σε αντιστάθισμα για τη συμφωνία αυτή. Υπάρχει μια κάποια ζώνη που δημιουργεί κάποια αμφιβολία για κάποιο τμήμα του στόλου. Είναι αλήθεια. Όμως παίρνουμε κάποια άλλα είδη. Λόγω αυτής της αλλαγής της ζώνης αλίευσης επιλύσαμε ταυτόχρονα και ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα της ε, αηφορίας των ε, αλλιευμάτων. Ήταν... Έχει συζητηθεί κατά κόρον ε, μέχρι το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πελαγικά είδη τα οποία θα, πρέπει να, θα πρέπει να προστατευτεί. Οι, σαρδίνες, οι σαρδέλες για παράδειγμα, που, η οποία έχει υπεραλιευθεί. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε την παραλίευση όπως το παρελθόν. Αλλάζοντας λοιπόν την αλλιευτική ζώνη, αυτόματα μειώνουμε την πίεση πάνω στα αλλιεύματα και μπορούμε να δεχθούμε αυτή την υψηλότερη ποσότητα. Κατά άλλα, ο κλάδος μας είπε ότι η κύρια προτεραιότητα είναι να έχουμε την μεγαλύτερη ποσότητα. Τους είπαμε ταυτόχρονα, θέλετε να συνεχίζετε να αλλιεύετε στην αρχική ζώνη, ζώνη, τότε θα πρέπει να μειώσουμε την ποσότητα και να έχουμε κάποια μείωση των ε, αλλιευμάτων του υποείδους των διαφόρων υποειδών ε, φρύσας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποδεχθούμε χωρίς ε, πληροφόρηση και συντονισμό, βλέποντας την προηγούμενη δραστηριότητα των αλληλευτικών στόλων, κατά 70% ήταν σε ζώνη που τώρα πλέον καθορίζεται από τους ε, Μαυρτανούς ως η νέα ελληνική ζώνη. Τώρα, κατά πόσον αυτό θα μπορούσε κάπως να αλλάξει, είναι προς εξέταση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αδιανόητο να ξαναγυρίσουμε στην αρχική αλληλευτική ζώνη. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εξάλλου, δεν είναι μόνο ότι τώρα έχουμε περισσότερα πελαγικά είδη με τα νέα είδη που υψέρχονται στη συμφωνία αυτή, αλλά έχουν και μεγαλύτερη αξία. Η αξία, δηλαδή η υψηλότερη αξία των νυχθείων είναι σχεδόν διπλάσια αυτή που θα έχουμε τώρα στη νέα αλληλευτική ζώνη σχέση με αυτή που είχαμε στο παρελθόν. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητήσαμε από το στόλο και απαιτεί από το στόλο να πάρει πολύ δυναμική άποψη το πώ προσεγγίζει την αγορά του. Αυτό βέβαια σημαίνει, δεν μπορεί να γίνει τσάμπα για τον στόλο, πρέπει να σκεφτούν δημιουργικά πώς θα εμπορευθούν τα νέα αυτά είδη στην αγορά. Και δεν μπορούμε να, το, να βλέπουμε μόνο, ε, αν θέλετε, κοντόφθαλμα μόνο ότι υπάρχει στο πρωτόκολλο, ό,τι υπάρχει στο πρωτόκολλο και τίποτα παραπέρα. Να το δούμε πολύ πιο ε, δημιουργικά και να ανταλλάξουμε, αν θέλετε, ότι τι αντιστάσεις θα δώσουμε σε σχέση με την αλλαγή της ε, αλληλευτικής ζώνης η οποία επέρχεται. Τώρα, η τρέχουσα, σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρήση, συνειδητοποιώ ότι κατά κάποιο τρόπο ε, είναι ατυχή σε στιγμή που είχε επιλεγεί. Καταρχά, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρχε ακόμα κάποια αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τι τεχνικέ συνθήκε και όρου. Η Μαυριτανία έπρεπε κάπω να το προσαρμόσει αυτό. Μετά μπήκαμε στα θέματα του βιολογικού κύκλου για τι γαρίδε. Πήκαμε στην περίοδο κλεισίματος, ε, του βιολογικού κλεισίματο, άρα δεν μπορούσαν να αλλιεύσουν ε, γαρίδες ούτω ή άλλω. Και για τα πελαγικά είδη παραδοσιακά αυτή είναι η εποχή με την χαμηλότερη δυνατότητα. Εάν λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορούν να αλλιεύσουν την ποσότητα που περιμέναν σε μια πολύ πιο περιορισμένη χρονική περίοδο, τότε είναι απόλυτα λογικό τώρα να είναι ακριβώ η περίοδο που δεν θα αλλιεύουν καθόλου. Ε, άλλωστε, η η, αυτή τη στιγμή, Μερλούκου και Τόνου είναι αυτοί που αλλιεύουν αυτή τη στιγμή. Τώρα ερχόμαστε στο κομμάτι που αφορά τα κεφαλόποδα. Εδώ και πάλι είναι το ερώτημα. Αγνοήσαμε τις επιστημονικές ε, συστάσεις. Κάθε άλλο, το αντίθετο. Βασιστήκαμε στις ε, πλέον πρόσφατες διαθέσιμες ε, επιστημονικές ε, πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια μας των διαπραγματεύσεων, το Ισπανικό Ινστιτούτο ήρθε με μια, μας προσθέσει μια μολέτη, την οποία είδαμε πολύ προσεκτικά, η οποία μελέτη αναφέρει ότι αν ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την διαχείριση των αλλιευμάτων, μπορούμε να προβλέψουμε πόσο και πάρα πολύ γρήγορα μπορούν να επανακάψουν τα αλλιεύματα. Και αυτό είναι αληθές. Ε, ένα αλίευμα που έχει απόθεμα με έναν κύκλο ζωής κάπου ένα-δύο χρόνια, σε συνάρτηση βέβαια με βιολογικές συνθήκες, όρους και σε συνδυασμό με τα μέτρα διαχείρισης τα οποία εισάγουμε, μπορούμε να έχουμε μια πολύ ευέλικτη ε, διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Αυτό το, θέξ, το θέξαμε το ζήτημα με τη Μαυριτανία και η Μαυριτανία αναγνώρισε ότι ενδεχομένως όντως μπορεί να υπάρξει πάρα πολύ γρήγορα ανάκτηση των ε, αποθεμάτων. Έχουμε άλλωστε σχετικές προφορίες που επιβεβαιώνουν ότι όντω είναι ένα αξιόπιστο σενάριο. Αλλά είπε επίση με Βρετανία ότι θα θέλαμε να δώσουμε στον στόλο την ευκαιρία να είναι ο πρώτος να αλλιεύσει αυτό το απόθεμα. Γιατί τα κεφαλόπεδα ε, ακριβώς είναι κάτι το οποίο ε, προσάδει προς τις αλλιευτικές ικανότητες των αλλιευμάτων μας. Ενώ δεν έχουν αντίστοιχα σκάφη ανοιχτή θαλάσση. Άρα θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το αλίευμα πρώτα για το στόλο μα και αν υπάρχει πλεόνασμα, τότε ναι, εσεί Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχετε την προτεραιότητα. Με αυτού του όρου, λοιπόν, ε, καταστρώσαμε τι σχετικέ ε, συνθήκε για τη σύναψη του πρωτοκόλλου αυτού που ευθυγραμμίζεται απόλυτα και με το διεθνέ δίκαιο. Δεν αρκεί να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κεφαλόπεδα πρέπει επίσης και τα παράκτια κράτη να αναφέρουν τι θέλουν να κάνουν με το απόθεμα αυτό. Εάν θέλουν καταρχάς να έχουν το δικαίωμα αλίευσης ε, των αποθεμάτων πρώτη, προφανώς έχουν αναφέρει το δικαίωμα. Ήταν και μια ιδέα που κυκλοφόρησε από τον κλάδο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή πάντα εμείς οι αλλιεύαμε, εμείς θα κρατήσουμε την προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι πολύ ισχυρό επιχείρημα. Εάν ο ντόπιο στόλο θέλει να, και έχει τη δυνατότητα να αλλιεύσει το απόθεμα αυτό, θα έχουν και την προτεραιότητα και αυτό έχουμε εισάγει στο πρωτοκόλλο αυτό. Υπάρχουν και πιο πρόσφατες πληροφορίες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση του αλλιεύματος. Τότε μπορούμε να αυξήσουμε τις ευκαιρίες που προβλέπει το πρωτόκολλο, μπορούμε να το συνεξετάσουμε με τη Μαυρετανία και είναι σίγουρο ότι αν υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα, εάν υπάρχει πλεόνασμα, τότε όντως μπορεί να είναι στη διάθεσή μας και αυτό πιστεύω ότι δεν θα παρουσιάζει κανένα πρόβλημα από καμία, κανένα πρόβλημα καμία όψη, ε, χωρίς να υπάρχει υπερβολική παρεμβολή και σύγκρουση μεταξύ του ντόπιου στόλου και του κοινοτικού. Και υπάρχει και απόλυτη αξιοπιστία, γιατί είναι ακριβώς ένα απόθεμα πολύ βραχαίος κύκλου ζωής, που μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Τώρα, το ερώτημα. Εάν θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε το πρωτόκολλο, τι πρέπει να κάνουμε. Το είπα, εάν οι νομικέ δυνατότητε, μα δίνουν δυνατότητα, να πούμε τώρα όχι και ξεκινάμε καινούργια παραδιαπραγμάτευση, υψέρχεται πρώτα μια νομική διάσταση, δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε σε κάτι πάρα πολύ γρήγορα, άρα αποκλείεται πλήρω η αλίευση, νομίζω ότι πρέπει να είναι απόλυτα σαφε αυτό, οι πάντε το καταλαβαίνουν. Και επίση, φανταστείτε τον ενθουσιασμό με τον οποίο το, η άλλη πλευρά θα αρχίσει η επαναδιαπραγμάτευση εάν το, το σχέδιο, το προτινόμενο τους απορριφθεί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα είναι και πάρα πολύ ανθουσιώδης και να πούν «Α, τώρα καταλάβαμε, σας δίνουμε όλα όσα θέλετε, παρακαλώ πολύ, ελάτε πάλι πίσω και κάντε ό,τι θέλετε». Είναι κατακλείδη, λοιπόν. Να, υπάρχουν και κάποια ε, συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα αναφέρω, αν θέλετε. Για παράδειγμα, έχουν, έχει απολυστεί κάπου 70% της ικανότητας αλίευσης γαρίδων. Αυτό είναι λάθος έχει ακουστεί. Απλώς υπήρξε επανακαθορισμός των ζωνών για την αλίευση των συγκεκριμένου στόλου. Ο μισός στόλος θα πρέπει να συνεχίζει και το έχουμε συσφαλίσει αυτό να εξακολουθεί να αλιεύει στις αρχικές ζώνες. Έγινε επανακαθορισμός της ζώνης για να μειωθεί η πίεση των, ε, των ε, μηχανότρατων ε, στο βάθο τη στον πυθμένα της θάλασσας και έχουμε εξασφαλίσει ακριβώ ότι θα, το μισό στόλο θα εξακολουθεί να αλλιεύει με τι προηγούμενε ε, συνθήκε και όρου. Άρα δεν μπορεί να κυκλοφορεί τέτοιο επιχείρημα. Αυτό λοιπόν το οποίο υποστηρίζουμε και ευχαρίστω να επισέλθω σε οποιαδήποτε τεχνική λεπτομέρεια θέλετε και σε εξέταση οποιοδήποτε επιχειρήματο θέλετε να μου αντιτάξετε. Λέω λοιπόν ότι αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την αλίευση, θα πρέπει να προχωρήσουμε, να δοκιμάσουμε, να δούμε ποιες είναι, τι μας φέρουν οι νέες τεχνικές συνθήκες και να επανέλθουμε να τις συζητήσουμε με τους Μαυριτανούς εάν το αλίευμα αναμονάδα και αναπροσπάθεια δεν είναι επαρκές. Κάτι άλλο σημαντικό σε ό,τι αφορά την, ε, σε ό,τι αν θέλετε, αν θέλετε την αντιπαροχή. Όταν η Μαυριτανία θα έχει τα χρήματα, τότε δεν πρέπει να φέρει καμία αντίρρηση. Είναι και ένα τέτοιο επιχείρημα το οποίο έχω ακούσει. Αλλά είναι εξαιρετικά υπεραπληστευμένη προσέγγιση στο θέμα. Καταρχά υπάρχει η ρήτρα καταγγελία. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά η ότι εάν μπορούμε να αποδείξουμε, αλλά βέβαια πρέπει πρώτα να υπάρξει η εφαρμογή του νέου αυτού πρωτοκόλλου, να πάει ο στόλος να λιεύσει και να δούμε συγκεκριμένα ε, τι γίνεται. Εάν δούμε λοιπόν ότι υπάρχει υποχρησιμοποίηση αυτή τη συμφωνία, μπορούμε να σταματήσουμε και την αντίστοιχη αντιπαροχή. Άρα δηλαδή δεν θα καταβάλουμε τα 70 ή μάλλον τα 67 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τα χάνουμε όλα τα χρήματα ευθύ εξ αρχή. Μπορούμε να τα καταβάλουμε και μετά να τα επαναδιακδικήσουμε είναι μια διαπραγμάτευση όπου η Μαυριτανία μπορεί να μα πει Αχ, τι ωραία, τώρα τα πήρα τα χρήματα, θα τα ξαναδίνω πίσω. Δεν είναι δυνατόν. Έχουμε μόνιμη σχέση με τη Μαυριτανία. Προφανώ πρέπει να σεβαστούν και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ. Και αν έχουμε ένα θεμητό ε, ε, δικαίωμα και αίτημα επιστροφή χρημάτων, μπορούμε να τα ζητήσουμε. Δεν είναι προ το συμφέρον των Μαυριτανών να πούν ότι Α, αν τα χρησιμοποιήσουμε καθόλου τη δυνατότητα αυτή, που είναι τελείως φανταστικό το σενάριο, τότε μπορούν να κρατήσουν 10-20 εκατομμύρια. Ναι, ή, ίσως, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα το έκαναν, γιατί θα διακινδύνευαν τη μελλοντική σχέση. Τέλος, γιατί δύο χρόνια ισχύω και όχι τρία, εμείς προτείναμε αρχικά να υπάρχει μια συμφωνία τριών ετών. Όταν όμως ε, προτάθηκαν οι διάφοροι χρηματοοικονομικές απαιτήσει, ήταν υπερβολικό πλέον το ποσό, γι' αυτό και φύγαμε από το τραπέζι διαπραγματεύσεων και γι' αυτό φτάσαμε τελικά στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο των δύο ετών, οπότε συμφώνησαν. Είπαν συμφωνούμε τις οικονομικές συνθήκες, ναι μεν το ποσό συγκεκριμένο το οποίο προτείναμε εμείς, αλλά μόνο για δύο χρόνια. Θεωρήσαμε ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης, γιατί έχουμε τουλάχιστον τεχνική δυνατότητα να συνεχίσουμε την αλίευση χωρίς να βρεθούμε εκτός για πολύ μακρά περίοδο. Ευχαρίστως παραμένω ανοιχτό για οποιαδήποτε εξέταση σε μεγαλύτερο τεχνικό επίπεδο, μεγαλύτερο βάθος όπως επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πολύ και ξαναδίνω τον λόγο στον εισηγητή. Όχι, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Έχω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Άκουσα με προσοχή. Και έχω την εντύπωση ότι εδώ λαμβάνουμε διαφορετικές πληροφορίες. Αυτά που μας είπατε τώρα στο τέλος θα ήθελα να τα έχω και γραπτά παρακαλώ για να τα διαβάσω με την ησυχία μου. Μπορείτε να μας τα δώσετε και γραπτός. Well, if you provide... για να στα δώσει όλα αυτά γραπτός γιατί το υπέρ θα ήταν μακροσκελέστατο το κείμενο. Ναι, το φοβόμουν, λέει ο κ. Δεπιπέρ. Ποια συγκεκριμένα σημεία αναφέρεστε. Ίσως, ναι, να το κάνουμε σε διμερές επίπεδο. Ναι, ο κ. Μάτα. Εν συντομία, γιατί πρέπει να επιστρέψω στην έδρα και να μοιράσω τον λιγοστό υπόλοιπο χρόνο. Ε, χαίρομαι που σχεδόν όλοι συμφωνούμε, ε, σχεδόν όλοι. Ε, συμφωνώ και, ε, και σε μεγάλο βαθμό και με την Σαβέλα. έχει αλλάξει η κατάσταση από το 2008 μέχρι σήμερα στα κεφαλόποδα για παράδειγμα. Είναι πολύ διαφορετική, είναι αλήθεια. Ε, ότι παλιότερα είχαμε υπερεκμετάλλευση, τώρα όχι. Τώρα μας λένε ότι έμεινε εκτός γιατί ανταγωνίζεται με τον Εθνικό Στόλο της Μαυριτανίας. Ε, καταλαβαίνω λοιπόν το επιχείρημα. Οπότε τι απομένει. Η, απομένει μόνο η δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούμε. Α, αυτό, αυτό στο οποίο είμαστε όλοι σύμφωνοι είναι το εξή. Το είπε ο κ. Δεπιπέρ. Στη Μαυριτανία δεν αρέσουν τα τεχνικά μέτρα, αλλά θέλει ε, συμφωνία. Και εμεί το ίδιο λέμε. Ε, ας ε, ξαναδιαπραγματευτούμε τα τεχνικά μέτρα. Προφανώ δεν είναι τόσο απλό. Γιατί μα λένε ή θα δεχτούμε αυτή τη συμφωνία ή θα μείνουμε ένα χρόνο χωρί αλεία. Χωρί αλίευση. Ε, για τι γαρίδε, ποιο είναι ο καλύτερο, Μήνα ο Αύγουστο που δεν τον χρησιμοποίησαν έτσι κι αλλιώ λοιπόν, πρακτικά αυτό έχει γίνει έτσι κι αλλιώ. για, τουλάχιστον για κάποιου στόλου. Δεν αλλιεύουμε. Από την άλλη μεριά, το βασικό πρόβλημα ενδεχομένω δεν είναι η αύξηση του κόστου. Οκ, okay, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό το βασικό κόστο. Ε, δεν είναι το, το βασικό πρόβλημα το κόστο για του στόλου. Αλλά τα προβλήματα δεν είναι, που είπα δεν είναι μόνο οικονομικά. Ε, ας πούμε ότι η αξία των αλλιευμάτων έχει αυξηθεί, δεν ξέρω πόσο. Σίγουρα όμως δεν έχει τριπλασιαστεί όπως τριπλασιάστηκε το κόστος των αδειών. Μετά, αυξάνονται οι τόνοι για τα πελαγικά είδη. Ωραία, αλλά μειώνεται η ε, επιφάνεια. Ε, Έχουμε διαφορετικά μίλια. Ναι, λέει ότι όμως τα, τα έχουν μεγαλύτερη ε, αξία. Δεν το ξέρω αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ειδοί για τα οποία γίνονται ε, υπάρχει, ε, υπάρχει ίδια τα οποία γίνεται υπεραλίευση όπως ενδεχομένως των πελαγικών ειδών αλλά δεν βλέπουμε να ζητάνε μείωση η Μαυριτανή. Τα κεφαλόποδα. Μπορεί να αναθεωρηθεί βέβαια η συμφωνία, λέει η Κομισιόν. Παράξενο. Ε, υπάρχει δυνατότητα νομικά, διατηρώντας ε, τα ε, δικαιώματα των εθνικών αλλιών κλπ. Το κείμενο όμως λέει με την αντίστοιχη προσαρμογή του αντιτίμου. το λέει αυτό η συμφωνία. Τα θετικά αυτής της συμφωνίας είναι ότι ε, κανένας δεν θα μας ανταγωνιστεί, λέει η Κομισιόν. Είδαμε όμως στην Αλία ε, IUU ε, πώ η Κομισιόν πράγματι <laughs> αναλαμβάνει να προστατεύσει τα συμφέροντα του κοινωνικού στόλου. Έχουμε χώρε οι οποίες δεν ε, είναι συνεργάσιμες και παρόλα αυτά δεν απαγορεύονται εισαγωγέ αλλιευμάτων αυτέ τις χώρε. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ότι ούτε εδώ ε, θα υλοποιηθούν αυτά τα καλά που υπόσχεται η Κομισιόν από τη Συμφωνία. Η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να το δοκιμάσουμε πρώτα, το δοκιμάσουμε πρώτα και μετά να την επαναδιαπραγματευτούν. Ε, εγώ λέω όχι. Τα 70 εκατομμύρια. Φοβάμαι ότι υπάρχει προηγούμενο. Ε, Κάποιοι άλλοι δεν μας υπέστρεψαν τα 70 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω αν οι Μαυριτανοί θα μας τα επιστρέψουν, θα δούμε. Μακάρι να γίνει και αυτό. Το πρωτόκολλο από οικονομικής πλευράς δεν είναι ε, ωφέλιμο. Ε, δημιουργεί προ... Ε, ζημίες και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ο αλευτικός κλάδος. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχουμε έξι ακόμα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό λοιπόν με τα χαράς δίνω πίσω το λόγο στον Πρόεδρο για να συνεχίσουμε. Ωραία. Αλλάζω καπέλο αλληλευτικέ Δυνατότητε και Οικονομική Ανυπεροχή προβλέπει η Συμφωνία Αλληλευτική Σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία του Μαυρικίου. Καλώ ορίζουμε και πάλι την Κομισιόν για να μα παρουσιάσει το καινούργιο πρωτόκολλο. Oui, merci, Monsieur le Président. Je, je reprends la... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παίρνω και πάλι το λόγο για να σας παρουσιάσω μια νέα συμφωνία, ένα νέο πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου. Πρόκειται για μια νέα συμφωνία και ένα νέο πρωτόκολλο. Λάβαμε μια εντολή διαπραγμάτευση από πλευρά του Συμβουλίου Φέτο τον Ιανουάριο και διαπραγματευτήκαμε αρχές του χρόνου. Ε, μονογραφήσαμε κάποια κείμενα με τον, τον Φεβρουάριο του 2012 με η νομοθετική πρόταση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 3 Αυγούστου. Πρόκειται λοιπόν, όπως έλεγα, για μια νέα συμφωνία και για ένα νέο πρωτόκολλο, με δεδομένο ότι η τρέχουσα συμφωνία ήταν αρκετά παλαιά, έπρεπε να επικαιροποιηθεί σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δει τις νέες προτάσεις για την μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής. Το τελευταίο πρωτόκολλο ε, έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2007. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή, αντικατοπτρίζει στην ε, δομή του τις προηγούμενες συμφωνίες που τις είχαμε διαπραγματευτεί από το 2004, δηλαδή καθορίζεται η αρχή, οι γενικές αρχές της εταιρική σχέσης, καθορίζεται η σχέση συνεργασίας ε, με επιστημονικά συμβούλια, θέτει τα διάφορα στοιχεία συνεργασία, την ε, μεικτή επιτροπή κλπ. Είναι ένα πλέγμα δηλαδή συνεργασία έτσι όπω το γνωρίζουμε. Η συμφωνία αυτή εταιρική σχέση συνήφθη για μια διάρκεια τριών ετών που θα είναι ένα ε, άριτος. Αναφέρεται επίσης ε, στο άρθρο 6 στην ε, ρήτρα αποκλειστικότητα. Έρχομαι στο πρωτόκολλο που είναι ένα λειτουργικό εργαλείο που καθορίζει δυνατότητες αλίευσης που πρόκειται δηλαδή για μια ε, συμφωνία ανατόνο και το πρωτόκολλο το οποίο ε, μονογραφήσαμε είναι μια διάρκεια τριών μηνών. Προβλέπει δυνατότητες αλίευσης, αλίας για 86 ελληνικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 41, ε, ε, μηχανότρατες και 45 ε, παραγάδια επιφωνίας. Η αρχική ποσότητα ήταν 5.500 τόνων και το οικονομικό αντιστάθμιο προβλέπεται είναι επίσης σχετικά μικρό. Είναι σε σχέση ακριβώς με την ποσότητα αναφοράς γιατί είναι ουσιαστικά 355.000 ευρώ για την πρόσβαση, συν 3.500 ευρώ ανά 302.500 ε, ε, ευρώ ε, ως βοήθεια. Άρα ένα σύνολο 660.000 ευρώ. Ε, είναι μια συμφωνία λοιπόν η οποία συμφωνεί με τι ε, συστάσεις του, της, στα πλαίσια τη Γενική Συμφωνία για την Αλία στον Ινδικό Ωκεανό. Γίνεται επίση αναφορά στην ε, αρχή ε, αποκλειστικότητας πέραν αυτή που έχουμε συμφωνία και έχουμε και διάφορα στοιχεία τα οποία λίγο πολύ μα δίνουν το σχεδιάγραμμα του, γενικού, του νέου πρωτοκόλου μετά την μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά την αρχή της αποκλειστικότητας, της αναλογικότητας, επικουρικότητας, ακόμα και μια ρήτρα η οποία έχει, ε, έχει ενταχθεί και αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια ρήτρα παραδείγματα σε ό,τι αφορά προβλέπεται να υπάρχουν 10 αλληλείς ε, της, ε, Χωτού Μαυρίκιου αν σκάφος. Ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία αφορούν την παρακολούθηση των σκαφών. Υπάρχει στοιχείο για την ε, μεγαλύτερη δυνατή απομάκρυνση, την μεγαλύτερη, την μεγαλύτερη δυνατή ακτή αλίας για τον ξένο στόλο, γιατί τα ευρωπαϊκά σκάφη επιτρέπεται να αλλιεύσουν σε απόσταση πέραν των 15 μιλίων από την παράκτη περιοχή του Μαυρικίου, ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιος ανταγωνισμός με τους Εντόπιου ε, αλείς μικρή κλίμακα. Ενδυναμώνεται επίσης η συνεργασία με το Μαυρίκιο σε περιφερειακό επίπεδο και επιτρέπει μεγαλύτερο σεβασμό και, και λήψη υπόψη του, των σχέσεων γενικά και των συμφωνιών ΑΚΕ. Επιμένω επίση το γεγονό ότι ότι στην ε, δημοκρατία του Μαυρικίου υπάρχουν και κάποιες, ε, κάποιες ε, μονάδες μεταπίεσης των ηχθείων που είναι πολύ σημαντικό γιατί, για την οικονομία της χώρας γιατί προσωπούν κάπου 6.000 θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου υπάρχει ιδέα και ένα κομμάτι του αλλιευτικού στόλου να συνεισφέρει στη λειτουργία της βιομηχανίας αυτής για την εκφόρταση και μεταπίεση των ηχθείων που είναι επιτόπου τόπου εγκαταστημένες. Αυτά σε ό,τι αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις καταστάσει, υποδομέ, ε, συγγνώμη, στο Δημοκρατία του Μαυρικίου, που είναι πολύ καλή ποιότητα. Ε, κλείνω εδώ σε διαφορά την αρχική παρουσίαση και παραμένω στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ενδεχόμενα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λόγο στον κύριο Σάντσε Πρεσέδο, τον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η συμφωνία δίνει συνέχεια σε σχέσεις οι οποίες ξεκίνησαν το 1989. Αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου πρωτοκόλου του 2007. Είναι μια στάνταρ συμφωνία που τηρεί τους κανόνες τέτοιων συμφωνιών σύμπραξης. Θα ήθελα να αναφερθώ στα εξή. Καταρχήν, η κατάσταση των αλλιευμάτων, των αποθεμάτων των αλλιευμάτων. Μιλάμε για την αλία τόνου. Η Επιτροπή Τόνου του, ε, του Ινδικού Ωκεανού ε, είναι υπεύθυνη. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη της για την κατάσταση των αποθεμάτων και αν το πρωτόκολλο ε, ευθυγραμμίζεται με, αυτήν, με αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Δεύτερον, θα ήθελα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τον ανταγωνισμό με τους ντόπιου αλείς. Οι ντόπιοι αλείς ε, νομίζω δεν ψαρεύουν τόνο, διότι ο τόνος αλίευεται σε μια ζώνη άνω των 15 μιλίων από τις ακτές, ενώ οι ντόπιοι αλείς ψαρεύουν στα 3 μίλια. Επίσης, οι ντόπιοι αλληλείς είναι 3.500 άτομα, από όσο γνωρίζω, και οι εργαζόμενοι ε, στις, ε, στη μεταποίηση του τόνου και σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες είναι 5.500 άτομα. Θα μπορούσατε λοιπόν να μου πείτε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα λιεύματα και δεύτερον ε, κατά πόσον οι δικέ μα αλλιευτικέ ε, δυνατότητε έρχονται σε αντίθεση, ή ανταγωνίζονται με τι αλλιευτικέ ε, την του Μαυρικίου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλει κάνει το λόγο? Όχι. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Κομισιόν θέλει το λόγο? Αν δεν σα είδα, έχετε το λόγο. Ε, αν μου επιτρέπετε, πολύ γρήγορα θα ήθελα να επανέλθω στα δύο αυτά σημεία τα οποία εθίγησαν. Λάβαμε υπόψη το σύνολο των ε, ε, μέτρων διαχείρισης για την περιφερειακό οργανισμό της Αλίας στην περιοχή του Ινδικού ωκεανού. Κύρια σημεία είναι που έχουν τεθεί σχετικά χαμηλό ποσοστό, που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό των ε, αλλιευμάτων στην περιοχή, έχουν καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις, ε, τα σχετικά λιτεύματα του είδους αυτού τόνου που είχαν παρατηρηθεί την εποχή δηλαδή που πριν από το 2007 προτού υπογραφεί το πρώτο πρωτόκολλο. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό με τους ντόπιου ε, το είπατε και ήθιος, παίρνουμε σαν αναφορά τα τρία μίλια. Πήραμε μια λοιπόν απόσταση 15 μιλίων από τις ακτές για απόσταση ε, ασφαλείας. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή εφαρμόσαμε την αρχή της ε, για να μην υπάρξει κανένας ούτε καν υποψία ανταγωνισμού με τους ντόπιου αλληλείς. Και ε, πρέπει να τονίσω ότι ούτω ή άλλω τα είναι τελείω διαφορετικά, γιατί από ό,τι ξέρουμε οι ντόπιοι αλλιεί ε, δεν στοχεύουν ε, στα είδη τα οποία προβλέπονται και καλύπτονται από το τρέχον πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Ωραία, περνάμε στο επόμενο σημείο. Αλληλευτικέ δυνατότητε και χρηματική αντιπαροχή, Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοκρατία τη Μαδαγασκάρη η Κομισιόν θα μας παρουσιάσει το καινούργιο πρωτόκολλο. Ο λόγος στην Κομισιόν. Yeah, merci Πάλι ευχαριστώ. Σε αυτήν την περίπτωση με τη Μαδαγασκάρη πρόκειται απλώς για μια ανανέωση ενός ε, πρωτόκολλου το, πρώτο είναι πρωτόκολλο εκπνέει στο τέλος του έτους και ήταν σημαντικό να υπάρξει ένα νέο πρωτόκολλο για να εξασφαλιστεί η συνέχεια στον ελευτικών δραστηριοτήτων. Η διαπραγμάτευση επίσης έλαβε χώρα αρχές του χρόνου. Τα κείμενα μονογράφησαν με τις αρχές της Μαδαγασκάρης στις 10 Μαΐου του τρέχοντος έτους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη υιοθέτησε τη νομοθετική πρόταση στι 19 Σεπτεμβρίου του τρέχοντο έτου. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρωτόκολλο που έχει μια διάρκεια δύο ετών και η διάρκεια αυτή εξηγείται από την ιδιαίτερη κατάσταση η οποία αντιμετωπίζει η δημοκρατία της Μαδαγασκάρης. Ξέρετε ότι είναι μια χώρα η οποία είναι σε μια κατάσταση πολιτικής μετάβασης αυτή τη στιγμή και ως εκ τούτου θεωρήσαμε κατάλληλο να, έχουμε, να προβλέψουμε μια διάρκεια του πρωτοκόλλου σχετικά περιορισμένη, ώστε να δοθεί δυνατότητα στον επόμενο πρόεδρο, στην επόμενη μας πολιτική εξουσία που θα προκύψει μετά τις εκλογές, που προβλέπονται κανονικά για τις αρχές του επόμενου έτους. Η νέα λοιπόν πολιτική ε, ηγεσία να ενδιαφερθεί για, το, για την αλία και να διαφερθεί για ένα νέο πρωτόκολλο. Παρά την πολιτική κατάσταση κάπως πολύπλοκη, την οποία έχουμε στο συγκεκριμένο νησί, παρόλα αυτά λάβαμε, κάθε δυνατή ε, με σχέση με τους συναδέλφους ε, εξωτερικής πολιτικής Πήραμε το πράσινο φω ότι με δεδομένο ότι βελτιώνεται η πολιτική κατάσταση μα είπαν ότι δεν μα εμπόδιζε τίποτα να υπογράψουμε ένα νέο πρωτόκολλο με τη Μαδαγασκάρη. Τώρα, το είναι, σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά τη αλληλεία του πρωτόκολλου αυτό, έχουμε 96 αλληλευτικά σκάφη, 40 ε, αθηναλιευτικά και 34 παραγαδιάρικα που ήδη μειώνονται σε σχέση με αυτό που είχαμε στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Απ' την άλλη αυξήσαμε κάπως ε, τη ε, χωρητικότητα αναφοράς στους 15.000 ε, τόνους από τους 13 για να λάβουμε υπόψη πραγματικά αλλιεύματα. Είναι μια μικρή προσαρμογή που δεν θα συνεισφέρει ουσιαστικά και δεν θα αυξήσει ουσιαστικά ε, την αλλιευτική προσπάθεια. Τώρα, η αντιπαροχή η οποία προβλέπεται είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατ' 950.000 ευρώ για την προσπέλαση και λίγο παραπάνω από 100.000 ευρώ για την ε, τομεακή υποστήριξη. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα τεχνικά στοιχεία που ίσως ενδιαφέρουν, ε, κάνουμε αναφορά στην, ε, σε κάποιες ε, υποχρεώσεις πάλι να υπάρχει ντόπιο αλληλευτικό πλήρωμα, 20 ουσιαστικά ε, ναύτες προσωπικό από τις χώρες ΑΚΕ και σε ό,τι αφορά την απόσταση, ε, την ε, υποχρέωση απόσταση από τις παράκτητε περιοχές, αυξήθηκαν σε 20.000 μίλια σε σχέση με 12 από την προηγούμενη συμφωνία. Από τον επόμενο χρόνο απαιτείται να τηρείται συστηματικά ηλεκτρονικό ημερολόγιο ε, του πλοίου για να παρακολουθούμε και την αλλιευτική δραστηριότητα και τα αλλιεύματα του στόλου σε σχέση με το πρωτόκολλο αυτή θα μπορούσαμε επίση να πούμε ότι τα επιστημονικά στοιχεία έγιναν σεβαστά. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο συνάδει στις καλύτερες ε, και πιο ε, ακριβείς και αυστηρές ε, οδηγίες. Και πάλι εδώ πέρα στοχεύουμε στον κυτρινόπλευτερο τόνο που δεν, που δεν κινδυνεύει στην περιοχή. Έχουμε επικαιροποίηση της συμφωνίας σε σχέση με τις ε, ε, συνθήκες που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση και τη συμφωνία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, είναι η ρήτρα της αναστολής ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ένα εχέγγυο. Η ρήτρα επίσης των όρων και της, και της αποκλειστικότητας, αλλά και σε ό,τι αφορά την περιφερειακή φύση αναφοράς του μηχανισμού. Οι προτάσεις μας ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις δίνουν μια αύξηση της αντιπαροχής που καταβάλλονται από τους εφοπλιστές κατά 25%, μια αύξηση της αντιπαροχής που καταβάλλονται από τους ε, κατόχους ε, ε, μηχανότρατας είναι 20%. Γενικό το τρόπο θα λέγαμε ότι η τομεακή βοήθεια που ε, επενδύθηκε στη Μαδαγασκάρη τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλίας και επομένως της καταπολέμησης της ε, λαθρέας αλίας και υπενθυμίζω ότι η Μαδαγασκάρη είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που αναγνωρίζεται στην περιοχή σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και επιτήρηση της αλίας. Γνωρίζετε ότι έχουμε χρηματοδοτήσει και χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα επιτήρησης στον Ινδικό ωκεανό που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και η Μαδαγασκάρη στον οργανισμό αυτό που επιτηρεί την ε, δραστηριότητα στον Ινδικό ε, ωκεανό, είναι ένας πολύ καλός ε, εταίρος και υποφελείται πολύ σωστά τα χρήματα τα οποία καταβάλουμε ως κομματική βοήθεια στα πλαίσια της δραστηριοτήτων αυτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο με τη Μαδαγασκάρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση συμφωνίας ε, εταιρικής σχέσης ε, αλίας ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαδαγασκάρης. Θα ήθελα όμως εντάχει να δείξω κάποια αμφισβητούμενα σημεία τα οποία θα ήθελα να σας επισημάνω. Θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε κατά κύριο λόγο να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση μιας υπεύθυνης πολιτικής αλλίας μια πολιτική υπεύθυνη αλλία, συγγνώμη, που θα λαμβάνει υπόψη και την ανάπτυξη τη χώρα αυτή, επιμένοντα ιδιαίτερα στα θέματα επιτήρηση τη αλλιευτική δραστηριότητα, πάνω στην σωστή διαχείριση των μέσων αλλία και στην βελτίωση των συνθήκων υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα αυτό. Αυτό το σημείο καθόλου δεν αναφέρεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω ότι θα μπορέσει να επανεξεταστεί η πρόταση αυτή και να συμπεριληφθεί ένα σημείο που θα αφορά τις ε, ε συνθήκες του τελικού προϊόντος. Τέλος, ό,τι αφορά την χρήση στα πλαίσια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, χρήση των οικονομικών ε, μέσων που διατίθενται από την Ευρώπη στον φορέα Μαλγκάς για την Αλία, θα πρέπει που, χρηματοδοτεί την εθνική πολιτική, είναι απαραίτητο να υπάρξουν αντίστοιχοι και εξωτερικοί χρηματοοικονομικοί έλεγχοι, ώστε να επαληθεύονται στις οποίες δηλώνουν. Πιστεύω ότι και αυτό το σημείο θα εμπλουτίσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως εκ τούτου ε, συμβουλεύω την ίδια την Επιτροπή αλλά και όλους τους συναδέλφους να σκεφτούν μια βελτίωση μιας ήδη πολύ καλής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις τροπολογίες που προτάθηκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που παρεμβαίνω ενώ ακόμα δεν έφτασα αλλά ήμουν αλλού. Ήθελα απλώς να πω ότι η συμφωνία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι θεμελιώδης για την ε, ε λειτουργία ε, ε, των, των ε, αλλιευτικών των, των αλλιευτικών που το 90% της φυριότητας το κάνουν εκεί. Οι ζώνες ορίζονται ε, αυστηρά, ώστε η Μαδαγασκάρη να έχει την εγγύηση ότι τα ύδατά της θα την χάνουν αϊφόρου και σωστής εκμετάλλευσης από τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Εξάλλου, η η χρηματοοικονομική βοήθεια, η αρρωγή προς τον κλάδο αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε. Και βέβαια τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας ήδη αναφέρθηκαν και είναι πολύ σημαντικός και ο έλεγχος με το ε, ηλεκτρονικό ημερολόγιο ε, καταστρώματος και με τα άλλα μέσα. Έχουμε μια αύξηση των αλλιευμάτων. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε ότι ταυτόχρονα υπάρχει και μεγαλύτερη χρηματική αντιπαροχή. Επίσης, ε, όλες αυτές οι αυξήσεις που έχουν προβλεφθεί των αλλιευμάτων είναι απόλυτα, ε, συμφωνούν απόλυτα με τα επιστημονικά ευρήματα και με όλα τα τελευταία ευρήματα, ώστε να υπάρχει μια συνοχή αν και της περιφερειακής οργάνωσης αλλίας και της σχετικής συμφωνίας. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη βεβαίως και τις ε, παρατηρήσεις του συναδέλφου κ. Ριβελίνη. Αυτό θα πω. Ευχαριστώ. Θέλει να προσθέσει κάτι η Κομισιόν. Ε, ναι, ευχαριστώ. Εντάχει, ευχαριστώ τους δύο βουλευτές για την συνεισφορά τους. Είναι αλήθεια ότι αυξάνεται η χρηματική αντιπαροχή στο πεδίο αυτό, πράγμα που θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε περισσότερες δράσεις ό,τι αφορά την επιτήρηση, τον έλεγχο, την ε, εξασφάλιση, την μεγαλύτερο έλεγχο σε ό,τι αφορά την υγιεινή των προϊόντων. Προφανώς δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο που έχουν πονομογραφεί όλα αυτά, γιατί απλώς έχουμε θέσει καταρχάς ένα πλαίσιο. Προβλέπεται όμως ότι τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύω του πρωτοκόλλου αυτού θα υπάρξει μια μεικτή επιτροπή η οποία θα συμφωνήσει πάνω στα συγκεκριμένα προγράμματα δράση και πώ θα γίνει καλύτερη δυνατή χρήση τη χρηματική αντιπαροχή για τον κλάδο αυτό. Μετά από διαπραγμάτευση ακριβώ και συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαδαγασκάρη. Άρα, τρει μήνε μετά την ε, λειτουργία του του πρωτοκόλλου αυτού θα έχουμε τις συγκεκριμένες δράσεις που αναφέρατε. Σε ό,τι αφορά το σημείο που θίξατε, να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο των δαπανών, θέλω να υπενθυμίσω ότι παρά την κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η Μαδαγασκάρη, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχει υιοθετηθεί ένα χάρτη ο οποίος ε, υλοποιείται και κάποια κονδύλια αναπτυξιακής βοήθειας που είχαν παγώσει πλέον έχουν ε, απελευθερωθεί. Άρα αρχίζει η εκταμίευση, αρχίζουν τα πράγματα πάντα πάλι να ε, ομαλοποιούνται. Αλλά προφανώς ε, είναι απαραίτητα κάποια μέτρα ε, δημοσιονομικού ελέγχου και ιδιαίτερα στα πλαίσια λειτουργία τη Μικτή Επιτροπής και χάρη ακριβώς των δομών μα και των επιτόπων αντιπροσωπιών μας μπορούμε να έχουμε έναν στενό έλεγχο των δαπανών που γίνονται εξ ονόματος του πρωτοκόλλου αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 14 διάφορα. Όπως σας είπα σήμερα το πρωί, θα κάνουμε μία ενημέρωση για την έκθεση Γκάλαχερ. Τεχνικά μέτρα. Κύριε Γκάλαχερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα τεχνικά μέτρα και η έκθεση για τα τεχνικά μέτρα που ενέκρινε η Επιτροπή πριν από μερικές εβδομάδες οδήγησαν σε ένα τριμερή διάλογο. Εσείς δυστυχώς δεν ήσασταν εκεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον Αντιπρόεδρο κύριο Στίβενσον που προέδρευσε. Η συνεδρίαση ήταν δύσκολη γιατί το χρονοδιάγραμμα ήταν μικρό και μας είπαν ότι δεν είχαμε αρκετό καιρό προετοιμασία για τον τριμερή διάλογο. Κάναμε λοιπόν ό,τι μπορούσαμε μέσα σε μια μισή ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας και για να είμαι ειλικρινής, είχαμε μεγαλύτερη πρόοδο τότε από ό,τι προηγουμένω σε όλη την προηγούμενη διαδικασία. Αναμένουμε ένα κείμενο. Το κείμενο όμως δεν περιείχε αυτά στα οποία είχαμε συμφωνήσει. Οι σκιώδεις εισηγητές τέθηκαν στη διάθεσή μας για μια συνάντηση. Απαντήσαμε επίσημα στο Συμβούλιο με τα έξι σημεία τα οποία θεωρούσαμε εμείς ότι μπορεί να είναι προβληματικά. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους το Σαββατοκυριακό. Τα δέχτηκαν αυτά που τους είπαμε. Και η Γραμματεία συμβούλευσε όλους τους κοιόδες εισηγητές για την κατάσταση και υποσχέθηκε να απαντήσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Δύο σημεία υπήρχαν τα οποία ήταν προβληματικά. Το, στα βόρεια της Σκοτίας, το αγγλοσκανδιναβικό τρίγωνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είπε πως είχε κάποιο πρόβλημα. Το Συμβούλιο όμως διαφώνησε. Τέλος, ένα άλλο σημείο, στο οποίο εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε συμφωνήσει, δεν έγινε όμως δεκτό στον τριμερή διάλογο, ήταν τα νέα και αναπτυσσόμενα είδη. Δεν έγινε δεκτός ο σχεδιασμός που προτείναμε. με την απάντηση ότι αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Αλλά περιμένουμε μία δήλωση στο τέλος του χρόνου έτσι μας είχαν πει, πέρασε αυτός ο χρόνος, δεν έγινε τίποτα. Όμως ελπίζω του χρόνου με την Ιρλανδική Προεδρία να έχουμε αυτή τη δήλωση. Να γίνει πρόοδος, διότι 12 μήνες πέρασαν και μείναμε στάσιμοι. Το κείμενο έφτασε στις υπηρεσίες μας εδώ, οι οποίες απάντησαν. Λογικά πρέπει να έχετε λάβει αντίγραφο διαφορετικά. Μέχρι τις 20 έως 21 Νοεμβρίου θα έχετε τα κείμενα στη διάθεσή σας. Εάν τα μέλη αυτή της Επιτροπής δεν είχαν εμπιστοσύνη στους κοιόδες εισηγητέ, δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε καθόλου. Και πιστεύω πως το ακούσαμε όλες τις απόψεις όλων των ομάδων του Κοινοβουλίου και πιστεύω πως αυτό φάνηκε, αλλά το Συμβούλιο προέβαλε εμπόδια και απειλές. Και νομίζω πως παίζει με τα νεύρα μας. Διότι πιστεύω πως αν αυτό είχε ε, αρχίσει από το Συμβούλιο αυτή η πρόταση, εμείς θα είχαμε λάβει υπόψη τι θέσει του, αλλά δεν έγινε έτσι. Και τέλο πάντων, να ευχαριστήσω, κλείνοντας την Επιτροπή, να ευχαριστήσω εσάς, Πρόεδρε, για την υποστήριξή σας, τους σκιώδεις εισηγητές για τη δουλειά τους διότι τώρα τα μικρά παράκτια σκάφη θα μπορούν να επικεντρωθούν στα είδη που πραγματικά θέλουν να αλλιεύσουν. Ευχαριστώ. Ε, δεν μου αρέσει πολύ να λέμε η καλύτερη δυνατή συμφωνία, αλλά σε αυτήν την περίπτωση νομίζω είναι μια καλή έκφραση. Θέλει κανεί το λόγο. Συμφωνούμε για το κείμενο. Ωραία. Η κυρία Λέβιν. Μάλιστα, θα ήθελα να σημειωθεί ότι ω συνήθω συζητούμε για αυτόν τον φάκελο και έχουμε πέντε δευτερόλεπτα να το κοιτάξουμε. Πριν συζητούσαμε επί ένα τέταρτο στην Επιτροπή για την έκθεση. Μετά έγιναν οι διαπραγματεύσεις και η συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Αλλά αμφιβάλλω αν όλοι πρόλαβαν να διαβάσουν όλα τα τεχνικά μέτρα δεν είχαν το χρόνο να κοιτάξουν τις συνέπειες όλων των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Και τώρα συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο αυτό. Δεν αμφιβάλλω ότι ήταν καλές οι προθέσεις των μελών που κατέθεσαν τις τροπολογίες, αλλά πολλές φορές αυτήν εδώ την Επιτροπή συζητούμε ότι πρέπει να έχουμε αξιολογήσεις ε, επιπτώσεων επιστημονικά στοιχεία χειροπιαστά και αυτό εδώ το έγγραφο να σας πω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις από τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι απαράδεκτο ότι πιεστήκαμε να το ξεφυλίσουμε έτσι στα γρήγορα και ως κοιόδες εισηγήτρια για τους πράσινους μου ήταν αδύνατο να κάνω τη δουλειά μου σε τόσο λίγο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν επιφυλάσσομαι για την στήριξη των πρασίνων για αυτό εδώ το έγγραφο, διότι δεν έγινε σοβα... η δουλειά σοβαρά, με σοβαρό τρόπο. Και δεν μπορούμε να κρίνουμε αν είναι βιώσιμο ή όχι. Αυτό. Κύριε Στίβενσον. Δεν πρόκειται να παρατείνω πάρα πολύ τη συζήτηση, αλλά πηγαίνοντας αυτά που είπε η κυρία Λόβεν, συζητηση αλλα πηγωντας αυτα που ειπε νομίζω ότι έγινε καταπληκτική δουλειά από τον εισηγητή. Εμείς θέλαμε την εισαγωγή και την ισχύ του πρώτου πρωτοκόλλου από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτου. Μα είπαν όμως αφέστατα ότι δεν θα υπήρχε χρόνος ούτε καν για, μια, για ένα δεύτερο γύρο τριμερού διαλόγου, προκειμένου να έχουμε και την, τα επίσημα μεταφρασμένα κείμενα για την ε, εφημερίδα. Συμφωνώ λοιπόν και ζητώ συγγνώμη για το ότι πιεστήκαμε, όντως και βιαστήκαμε, αλλά παρόλα αυτά, έχοντας αντιμετωπίσει και το Κοινοβούλιο στον τριμερή διάλογο, παρόλα αυτά φτάσαμε σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο προσπάθησε να παραμείνει ε, αμετάβλητο στη θέση του κατά διάρκεια διαπραγμάτευση μέχρι ότου πάσαμε, αν θέλετε, και είχαμε πλέον άτυπε συζητήσει και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε στη συμφωνία και ιδιαίτερα σε κάποια ε, θέματα τα οποία ήταν εξαιρετικά κρίσιμα και που θα ήταν προ όφελο όχι μόνο για τη διατήρηση των αλλιευμάτων, αλλά και υπέρ των αλλιέων. Νομίζω ότι ναι, ήταν βιαστική δουλειά, όμω παρόλα αυτά ήταν μια δουλειά την οποία χειρίστηκε πάρα πολύ καλά ο εισηγητή και αξίζει τα συγχαρητήριά μα. Ωραία. Επίσης τα διάφορα, ε, ήταν απόφαση των συντονιστών, αλλά να το γνωρίζετε κι εσείς, ε, σήμερα το πρωί για τις αντιπροσωπείες του, του επόμενου έτους ε, είχαμε, είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την αποστολή στα Κανάρια επειδή συμπίπτει με το καρναβάλι. Οπότε τέθη το θέμα του να ε, αλλάξει η με τη Δανία με την Ιρλανδία. Όμως άλλες πρόσθετες δυσκολίες ε, με τη φιλοξενούσα ε, ε, με τον φιλοξενούντα στην Δανία που δεν θα είναι παρόν εκείνη την εποχή κατέστη αδύνατον να πάμε στην Δανία αντί να πάμε στα Κανάρια. Ε, προς το παρόν εκκρεμεί. Θα ξαναγίνει μια συζήτηση με τους συντονιστές ε, να δούμε μήπως βρούμε μια άλλη ημερομηνία. Και ηλεκτρονικά σας ενημερώνουμε και παίρνουμε την απόφαση σαν να είχε ληφθεί σήμερα. Σαν να είχε ληφθεί σήμερα. Σε ό,τι αφορά τι ανακοινώσει του Πρόεδρου σχετικά με τι αποφάσει των συντονιστών, σα ε, είπα ποιο ήταν το βασικό θέμα. Δεν ξέρω αν εσεί έχετε οτιδήποτε άλλο. Μα το... Ε, μας γράφετε ένα email και το λαμβάνουμε υπόψη. Προσεχή συνεδρίαση 28 Νοεμβρίου το πρωί και το απόγευμα και 29 Νοεμβρίου μόνο το πρωί. Αν δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. finished Thank you. Thank you, Ah,